Καθίστε παρακαλώ. Λοιπόν, ε, σχετικά με το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, πρόκειται για την υιοθέτηση της ημερησίας διάταξης. Υποθέτω ότι συμφωνείτε όλοι και το επόμενο θέμα είναι η η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 16ης Ιουλίου 2009 που δεν ακούω ούτε εκεί κανένα σχόλιο. Το τρίτο θέμα είναι η ανακοίνωση της Προέδρου ότι και πάλι σήμερα υπάρχει ε, ε, web streaming οπότε παρακαλώ να είσαστε ε, προσεκτικοί και Ερχόμαστε στο 4, έγκριση του σχεδίου χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της Επιτροπής ΕΚΟΝ για το 2010. Αυτό είναι το ίδιο ε, εκτός από τους συντονιστές για τις ε, 24 Ιουλίου στις 23 ε, το απόγευμα δεν είναι δυνατόν να έχουμε συνεδρίαση διότι συμπίπτει με άλλες συνεδριάσεις αλλά όπως είπα και προηγουμένως ε, έχουμε έχουμε ε, προβλέψει πολλές συνεδριάσεις για του χρόνου διότι θα έχουμε φόρτο εργασιών. Λοιπόν, Εάν ε, συμφωνείτε θα θεωρήσουμε ότι έχει υιοθετηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και τώρα έρχομαι στην ανταλλαγή απόψεων με το Sir David Tweedy, πρόεδρο του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τον οποίο καλωσορίζω εδώ. Την τελευταία φορά που που συναντηθήκαμε ήταν τον Απρίλιο του 2007. Οπότε τώρα επί 15 λεπτά θα μας παρουσιάσετε ε, τα λογιστικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε, ιδίω όσον αφορά το IIS 39 και το USFASP και ενδεχομένως μπορείτε να μας πείτε και για τα θέματα της συνάντησης των G20. Ξέρω ότι είναι πολλά θέματα. Έχουμε ένα έγγραφο που αναφέρεται εις ε, την ε, ε, ομιλία το οποίο θα σας διανεμηθεί και ε, μας δίνονται έτσι διάφορες γενικές παρατηρήσεις μετά όταν τελειώσει, αφού τελειώσει λοιπόν ο κύριος ε, Τουίγκλ θα, θα έχουμε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ να ξαναέρθω και να συζητήσουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσεως θα αναφερθώ στην οικονομική κρίση παρόλο που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη αλλά αν έχετε και σε άλλα θέματα ερωτήσεις ε, θα απαντήσω ευχαρίστως. Ένας πολυεκατομμυριούχος λοιπόν ε, κεράτησε, κάλεσε φίλους του εις ε, το το, τους έδειξε μία, ε, τους κάτσε στην πισίνα του γεμάτη κροκόδιλους ε, και ε, του πρόσφερε 10 εκατομμύρια δολάρια να παντρευτούν την κόρη τους και ούτε καθεξής. όταν λοιπόν βγήκε ο πρώτος του λέει τι θέλεις παρανοπόλα όλα λέει να βρω αυτόν που με έσπρωξε γιατί πήδηξε κάποιος αμέσως μέσα. Λοιπόν, ε, τώρα βρισκόμαστε στο σημείο πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, διότι πρόκειται για ένα κρίσιμο θέμα για τον κόσμο και για την Ευρώπη και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε την οικονομική μας υποδομή ε, ε, πρέπει να έχουμε μία αμφίδρομη συνεργασία και σε αν χρειάζεστε ε, σε μία ερώτηση μπορείτε να την αναφέρετε κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου χωρίς να περιμένετε να τελειώσω υπήρχαν ορισμένα λογιστικά πρότυπα ένα θέμα το οποίο, για το οποίο πρέπει να είναι πολύ περήφανη η Ευρώπη διότι η Ευρώπη ήταν αυτή η οποία πρώτη παρουσίασε τα λογιστικά πρότυπα το 2001-2002 τα οποία υιοθετήθηκαν από διάφορες χώρες τώρα 117 τις έχουν υιοθετήσει ακόμη και η Κίνα προσχώρησε το 2007 πέρυσι ήταν το Ισραήλ, φέτος ήταν η Χιλή ε, και το 2010 θα είναι η Βραζιλία, το 2011 η Κορέα, η Ινδία, η Ιαπωνία, ε, μετά το Μεξικό, δηλαδή ε, σιγά σιγά προσχωρούν όλο και περισσότερες χώρες και το Ηνωμένε Πολιτείε ακόμη δεν έχουν προσχωρήσει γι' αυτό και προσπαθούμε να ε, εξασφαλίσουμε ότι τα αμερικανικά από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ε, δεν θα διαφέρουν πολύ ώστε σιγά σιγά να αναγνωριστούν διεθνώς και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα θα σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητές μας. Αυτό προφανώς ε, ε, χρειάζεται. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι στις Ηνωμένε Πολιτείε, την επόμενη εις ε, την η Ιαπωνία και το ΕΚΟΦΗΝ θα συνέλθει σε ένα μήνα περίπου και έχω λάβει την επιστολή που έστειλε προς τα μέλη ε, ο πρόεδρος εν ώψη των ε, G20 αναφέροντας τα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη. Θέλουμε να εξετάσουμε ε, διάφορα θέματα, δηλαδή προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε διάφορα θέματα, να έχουμε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα ε, συμβουλευτικό συμβούλιο ε, στο οποίο πολλοί ε, προέρχονται από την Ευρώπη ο Στίβεν Χάιντρο Γενικός Διευθυντής από τον Οργανισμό Ασφαλίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ε, ένας Γάλλος, ένας υπουργός οικονομικών της Ιταλίας, ο Χάνς Πίτερ Μίλλερ, ο Λουκάς Παπαδήμας, ο αντιπρόεδρος της ε, ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξέδωσαν μία έκθεση τον Ιούλιο την οποία ευχαρίστως θα σας διαθέσω και έκαναν διάφορες συστάσεις ε, για σας αυτά ίσως σας φαίνονται ε, απόμακρα αλλά εγώ όταν πήγα σε μια εταιρεία ε, λογιστών είχα μαζί μου δύο συναδέλφους από το Λονδίνο οι οποίοι ήθελαν να ενημερώνονται και όταν όταν ε, ε, ε, πήγαν στο, στην εφημεριδοπόλη τους είπε θέλετε τη σημερινή ή τη χθεσινή λέει τη σημερινή τότε θα έρθετε αύριο Λοιπόν, ε, αυτό τους εξέπληξε πάρα πολύ, διότι ε, από τα θέματα που ενδιαφέρουν υπάρχει αξία και ρευστότητα στην αγορά, να ε, υπάρχει εξασφάλιση και ειδικευμένοι μηχανισμοί και αποκάλυψη του κινδύνου όσον αφορά καταρχήν τη ρευστότητα της αγοράς η οργάνωσή μας πέρυσι είχε δημοσιεύσει μία έκθεση. Βεβαίως ενδέχεται να διαφέρουν οι απόψεις μας από τις Αμερικάνικες και γι' αυτό προσπαθήσαμε να συγχωνεύσουμε τις δύο προτάσεις και ε, να ε, τα ενσωματώσουμε στα λογιστικά μας πρότυπα τα οποία θα δημοσιευθούν του χρόνου. Επίσης θέλουμε διαφάνεια για να ξέρετε τι κίνδυνος υπάρχει σε τέτοια κρίση και επίσης πολλές εταιρείες οι οποίες ε, μέχρι τώρα χρησιμοποιούν τα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα τώρα χρησιμοποιούν τα ε, διεθνή. Ε, ε, βεβαίως εξαρτάται αν πρόκειται για θηγατρικές αμερικανικών εταιριών οπότε ακολουθούν την αμερικάνικα και προσπαθούμε να τις θυμώξουμε ακόμη περισσότερο το βασικό μας θέμα είναι ε, τα, τα πρότυπα που ονομάζονται IIS 39. Βεβαίω είναι κάτι ίσως το ακατανόητο. Εμείς το, το έχουμε κληρονομήσει και το κληρονομήσετε και εσείς. Παρ' όλα αυτά όμως εξετάσαμε τα διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει ε, κατά την ε, εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών ε, ζητήθηκαν διευκρινήσεις γιατί οι κανόνες διαφέρουν από τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ε, επίσης ε, ο καθορισμός της σωστής αξίας όταν πρόκειται για χρεόγραφα τα οποία είναι προς πώληση και να μην υπάρχουν παρανοήσεις εάν θέλετε να τα αποσύρετε. Όσον αφορά τις μη αγορές καθορίσαμε την την, ε, τις αρχές μας και ε, όσον αφορά τα εμπόδια ε, είναι το θέμα στο οποίο το Συμβούλιο Υπουργών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησαν να δράσουμε και προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε το IS 39 και να εκδώσουμε ε, τα στοιχεία μέχρι το τέλος του χρόνου. Ε, θέλουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε μία πρόταση σχετικά με αυτά τα νέα, ε, νέα πρότυπα ε, πράγμα το οποίο έγινε και στο G20 μας συνεχάρισαν πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα κοίταξαν. Τον Απρίλιο ε, τα πρότυπα αυτά αναφέρθηκαν στα εμπόδια που δημιουργούν ορισμένες καταστάσεις για να επιταχύνουμε την προσέγγιση μας ε, και την 1η Απριλίου ζητήσαμε να υπάρχει ίση μεταχείριση στην αγορά ε, διότι αν θέλουμε να μειώσουμε τα πρότυπα πρέπει να βελτιώσουμε τα πρότυπα. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τα πρότυπα που αναφέρονται σε αυτά τα εμπόδια και τις αδυναμίες. Στη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ τον Ιούνιο υποσχέθηκα ότι θα έχουμε ολοκληρώσει την αναθεώρηση μέχρι το τέλος του χρόνου και νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Θα μπορέσουμε λοιπόν να εξετάσουμε ε, τα θέματα των εμποδίων και της ανακατατάξεως που μας ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε σχόλια από 200 άτομα. Συναντήσαμε 70 θεσμικά όργανα και τράπεζες ε, ε, ασφαλιστικές σημαντικές εταιρείε οι οποίες ασχολούνται με τέτοια θέματα. Έχουν υπάρξει και άλλες ε, συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι εγκαίρως. Ε, πρέπει να είναι έτοιμο το σύνολο των προτάσεων να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο για να διευκολύνουμε τη διαδικασία και θα ήθελα εδώ να προτείνω ορισμένα θέματα τα οποία θεωρώ πιο σημαντικά. Πρώτον, η πρότασή μας θα μειώσει σημαντικά το, την περιπλοκή της ε, ε οικονομικής λογιστικής. Δεύτερον, ε, οι προτάσεις μας ε, είναι, συνάδουν με ε, τις, τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων και ιδίως της Επιτροπής της Βασιλείας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική πραγματικότητα και να υπάρχει διαφάνεια θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει ορισμένα θέματα να παρουσιάζονται σε βάση κόστους και πια σε σημερινή αξία δεν νομίζουμε ότι ε, οι τράπεζες πρέπει να αξιολογούνται βάσει της ε, δίκαιας αξίας και ε, εάν θέλουμε να δείξουν, αν θέλουν να δώσουν δάνεια θα πρέπει να παρουσιάζουν το κόστος και αυτοί οι οποίοι αγοράζουν με το τοχές τοξικά θέματα όλοι αυτοί με τα λεγόμενα ε, στοιχεία προσπαθούν να παρουσιάσουν την, ε, ε, την δίκαια τιμή. Θέλουμε όμως να καλύψουμε τις ανάγκες των ενδιαφερομένων θεσμικών οργάνων και να προλάβουμε θέματα που δεν μας έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά τα οποία θα ε, προκύψουν και θα πρέπει να καταταγούν στα στοιχεία του κόστους. Να υπάρξει μία ανακατάσταξη της ε, εναλλακτικής λύσης ε, δίκαιας αξίας σε άλλες κατηγορίες και ε, να υπάρχουν αλλαγές στις ανάγκες ε, υποβολής στοιχείων ορισμένοι μας ε, είπαν ότι χρειαζόμαστε περισσότερα, περισσότερο χρόνο. Εάν όμως δεν είμαστε έτοιμοι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να υιοθετήσουμε τα αμερικάνικα πρότυπα και ε, η Επιτροπή μας δεν ήθελε ε, να κλείνει προς τα αμερικανικά πρότυπα διότι προλίγων ετών χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο αυτή για τις εκθέσεις τμήματων και δεν πιστεύουμε ότι εδώ τα αμερικάνικα πρότυπα είναι η λύση. Ακόμη και αν δεχθούμε τις αμερικανικές προτάσεις δεν θα υπάρχει ισοτιμία διότι έχουμε διαφορετικούς κανόνες, διαφορετικά εμπόδια και ε, ε, τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην Αμερική προκαλούν διαφορετικές αντιδράσεις άρα διαφέρει η νομοθεσία μας στο θέμα αυτό μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Επίσης ε, οι προτάσεις δεν είναι κάτι που διατυπώθηκε σε λίγους μήνες. Ξεκινήσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2007. Πέρυσι δημοσιεύσαμε ένα έγγραφο συζητήσεως σχετικά με τις προτάσεις αυτές, άρα δεν πρόκειται για νέα στοιχεία. Επιπλέον, πέραν της προτεραιότητας αυτής, ε, εξετάσαμε ε, ένα άλλο θέμα που μας ζήτησαν το G20 σχετικά με τις διατάξεις για δανειοδοτήσεις. Ε, και να μην χρησιμοποιούμε το τωρινό, για να μην χρησιμοποιούμε την τωρινή ε, μέθοδο για τις ζημίες και να καλύψουμε και το hedging μέχρι το τέλος του χρόνου. Χρειάζεται διαβούλευση. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι επιτροπές ε, όπως αυτή ε, και οι τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν αυτά τα θέματα και θέλω να ε, διασφαλίσω όλους ότι στο λίγο χρόνο τον οποίο είχα περιορίστηκα μόνο σε θέματα τα οποία έχουν σχέση της, ε, με την οικονομική κρίση αλλά έχουμε άλλα θέματα πολύ σημαντικά και τα οποία επεξεργαζόμαστε μαζί με την Αμερική για να διατυπώσουμε κοινά πρότυπα για τις συντάξεις, για την ασφάλεια, για τις συμβάσεις και ελπίζουμε ότι η εργασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί ως το 2011. Θα σας ενημερώσουμε ε, για το πώς προχωράμε και αν ε, έχουμε κάποια ανησυχία θα έρθουμε να συζητήσουμε μαζί σας είτε στην Ολομέλεια είτε σε μικρότερη ε, επιτροπή για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Ε, θα πρέπει η Ευρώπη να μας στηρίξει σε αυτό το πολύ ουσιαστικό θέμα. Είστε ένας ε, βασικός μας στυλοβάτης και χαιρόμαστε γι' αυτό διότι είναι η καλύτερη ευκαιρία την οποία έχουμε ε, να έχουμε ε, συνολικά πρότυπα. Έπαιζα παιδόσφαιρο όταν πήγαινα σχολείο και θυμάμαι ότι μία μέρα κάποιος χτύπησε την ε, μπάλα και δεν πρόλαβα ούτε να τη δω. Τη δεύτερη φορά όμως είχα είχα αντιδράσει γρήγορα διότι ουσιαστικά ακόμη αντιδρούσα στην πρώτη, στο πρώτο χτύπημα. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει και εδώ αλλά να καταλήξουμε γρήγορα σε συνολικά πρότυπα ώστε να είμαστε όλοι καλυμμένοι. Ευχαριστώ. Right. Ευχαριστώ πολύ. Είχε σβήσει το μικρόφωνο μου. Μας μαλώνουν όταν χρησιμοποιούμε λάθος μικρόφωνο εδώ. Αυτό το πρόβλημα έχουμε. Πρώτος στον κατάλογο των αγοριτών, jean Jean-Paul Gauzes. Θα πρέπει να αλλάξετε εδώ το κουμπάκι σας στα ακουστικά για να ακούτε γαλλικά. Να πάτε στο νούμερο 3. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε να μας δώσετε πληροφορίες. Θα είμαι ευθύ. Αναφερθήκατε στα διάφορα θέματα στη, σύνολη, στη σύντομη επισκόπησή σας. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Μικρές ερωτήσεις, μικρές το δέμα, αλλά σημαντικές. Πώς θα ενσωματώσετε τις συστάσεις του G20 στις ε, πρόσφατες προτάσεις τις πρόσφατες προτάσεις του G20, στις προτάσεις σας. Δεύτερον, κάτι που αναφέρατε, αλλά είναι σημαντικό θέμα, έδειξε η κρίση ότι σε μερικές περιπτώσεις ε, δεν ήταν αρκετά κάποια μέσα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα, διότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Και σχεδιάζετε να λάβετε υπόψη σας την ε, θεμελιώδη αρχή της Επιτροπής της Βασιλείας τι συστάσει Επιτροπή τη Βασιλεία που μέχρι τώρα ε, έχουν αγνοηθεί βασικά. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία ερωτήματά μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Οι προτάσεις των G20 ταιριάζουν με αυτά που προτείνουμε. Θέλουμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα, να έχουμε παγκόσμιε προδιαγραφέ και την περασμένη εβδομάδα μάλιστα προσπαθήσαμε να ολοκληρώσουμε αυτέ τι εργασίε, το πρόγραμμα με τις ΣΥΠΑ μέχρι τον Ιούνιο 2011. Όλα ταιριάζουν με τι προτάσει των G20. Η τίμη αξία, η δίκαιη αξία, το fair value κάποια στιγμή δεν δούλεψε σωστά. Τι είδαμε από την κρίση. Λοιπόν, ότι η οικονομική κρίση, η Βουλευτική Επιτροπή την οικονομική κρίση μας είπε ότι οι λογιστικοί υπολογισμοί υποτίμησαν τις απώλειες διαφορών θεσμών. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει τόσο θεμητή προσέγγιση στα λογιστικά όπως ε, υπολογίζεται στη ΣΥΠΑ. Είδαμε ότι οι τράπεζες κατά μέσο όρο είχαν 25% στοιχεία ενεργητικού στο fair value. Ε, τα προβλήματα ήταν στις δανειοδοσίες. Εκεί ε, υπέστησαν τις απώλειες. Είναι έχουν υποτιμηθεί αρκετές fair value, αλλά οι απώλειες υποτιμήθηκαν και δεν καλύφθηκαν πλήρως ή αρκετά γρήγορα. Όσον αφορά τώρα τι συστάσει Επιτροπή τη Βασιλείας, ε, νομίζω ότι ταιριάζουμε αυτά που μα είπε η Βασιλεία. Δεν διαφωνούμε τη Βασιλεία. Οι ε, δείχνουν ότι οι δανειοδοσίε είναι σωστέ. Αν κινηθεί κανεί επί τη βάση ανάκτηση των τόκων, και να ανακτήσει το κεφάλαιό σου, τότε όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Τώρα, εκεί που υπάρχει είναι απρόβλεπε οι ροέ του ρευστού, το συζητήσουμε και το συζητούμε και με την Επιτροπή της σταθερή Αξίας. Θα το συναντήσουμε τις επόμενες εβδομάδε. εβδομάδες. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ ημών και βασιλεία. Ευχαριστώ. Ε, Επόμενος είναι ο Μπάλτς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σε David, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί για άλλη μια φορά το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον τονίσατε ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι φυσικά στο μέλλον θα πρέπει να σας υποστηρίξουμε και θα σας υποστηρίξουμε σίγουρα. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτο, από το board η προτινόμενη μείωση της, ε, των κατηγοριών αξιολόγησης ουσιαστικά από όλους τους ειδήμονες θεωρείται ως συνεισφορά για την απλούστευση των περίπλοκων και σύνθετων διατάξεων. Από την άλλη πλευρά οι διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με το fair value και το amortized costs αποκλειστικά με βάση τις συγκεκριμένες ιδιότητες των επιμέρους ομολόγων θα πρέπει να γίνεται. Εσείς πώς κρίνετε την πρόταση οι υποχρεώσεις αυτές να προσανατολίζονται σε σχέση με πρότυπα επαγγελματικά ώστε οι επιχειρήσεις την στρατηγική τους όσον αφορά τέτοιου είδου κριτήρια που θα πρέπει να τα προσαρμόζουν ή να τα σταθμίζουν. Μια δεύτερη ερώτηση. Ασκήθηκαν επικρίσεις ότι οι προτάσεις του Board για την αξιολόγηση των μέσων ιδίου κεφαλαίου δεν οδηγεί σε διαχωριστικές σαφείς γραμμές σε σχέση με τα καθαρά κέρδη και τις απώλειες. Αυτό θεωρείται μια μη ενδεδειγμένη μορφή ισολογισμού και αν για παράδειγμα έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική που ακολουθούμε, που παρακολουθούμε, που μπορεί να έχει ενδιαφέρουσες πτυχές γι' αυτό, εσείς πώς κρίνετε αυτά τα επιχειρήματα και τι έχετε να θέσετε ενώπιον αυτών. Ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα Έχουμε τέσσερις κατηγορίες με τους παρόντες κανόνες και δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Ένα είναι εύκολο, αν εμπορεύεσαι από αγορά σε αγορά, υπάρχουν κέρδη και απόλυση όσον αφορά το εισόδημα. Αδιαμφισβήτητο αυτό. Μετά, αν κρατήσει κάτι μέχρι ότου οριμάσει, δεν σε ενδιαφέρουν οι αλλαγέ τη αξία του. Οπότε είναι μια κατηγορία αξιογράφων που κρατούνται για να οριμάσουν. Και μετά υπάρχει μια επώνυα. Ίσως κάποιοι θεσμικοί φορείς κρατούν κάποια πράγματα σε αυτή την κατηγορία, αλλά αν χρειαστούν κέρδη και υπήρχε κέρδο για κάποιο αξιόγραφο, μπορεί να τα πουλούσαν για να αυξήσουν τα κέρδη. Αυτό πλην κληρονομήσουμε αυτέ τι προδιαγραφέ. Οι επιχειρήσει θεώρησαν ότι αυτό ήταν άδικο. Δηλαδή, αν πουλούσαν, έπρεπε να τα διαθέσουν όλα στην αγορά και να μπουν σε άλλη κατηγορία. Και αφήβραν τρίτη κατηγορία προ πώληση. Και αυτή η κατηγορία ήταν το πρόβλημα που είχαμε όσον αφορά του υπολογισμού και τι αναφορέ. Πολλά, πολλά στοιχεία που θα ήταν προσωριμότητα πήγαιναν στη διαθεσιμότητα προσπόληση πώληση, διότι υπήρχαν ε, σημαδευόταν αν θέλετε κάποια αξιόγραφα αν τα κρατούσε κανείς προσωρίμανση. Διαθέσιμα προσπόληση πώληση αυτή η κατηγορία πήγαιναν προς αγορά. Τα κέρδη και οι δεν ελαμβάνονται υπόψη στα για τα κέρδη μέχρι ότου να γίνει πωλήση και δεν μπορεί να μεταφέρει τι απώλειες στους υπολογισμούς και για, γι' αυτό φέραμε κανόνες λέγοντας πώς δείχνει κανείς ότι οι απώλειε ήταν μόνιμες και αυτές ήταν οι κανόνες περί δυσχεριών για χρεόγραφα δείχνεις τιμή μόνιμη fair value μπορούσαν να την αποσβέσεις για άλλα ομόλογα έδειχνε στις βλάβες όταν ήταν σημαντικές οι απώλειες στον αφορά το ομόλογο ή παρατεταμένες και δεν ήταν αντιστρεπτές οι συνέπειες. Αυτοί ήταν οι κανόνες, οι αμερικανικοί κανόνες. Πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι γελίο. Έχουμε τρεις διαφορετικούς κανόνες για απώλειες σε μια προδιαγραφή. Μπορούμε να καταλήξουμε με ένα νέο κανόνα για αξιόγραφα που κοστίζουν και θα χαθούν και όλοι οι περιορισμοί όσον αφορά τι μπορεί να συμπεριλάβει στο κόστος. Αυτά που ήταν προς πώληση θα προχωρήσουν προς τα κάτω όσον αφορά τη σειρά στα προς πώληση. Δίκαιο, διότι όταν εμπορεύεσαι θα έπρεπε να, να υπάρχει κάποια αξία αν δανειοδοτείς και συλλέγει τόκου, αυτέ είναι οι χρηματικέ ροέ που πρέπει να αντικατοπτρίζονται και αυτή είναι η κατηγορία κόστου. Έπρεπε να μπουν σε αυτή την κατηγορία. Τώρα οι μακροχρόνιε απώλειε και τα κέρδη, ξέρουμε αυτό το θέμα. Είναι γεγονό ότι ένα σημαντικό τομέα είναι οι ασφάλειε Επί του παρόντος συνομιλούμε με αυτό το τομέα επικοδομητικά για να ετοιμάσουμε νέα προδιαγραφή που θα προσμετρά τις ευθύνες όσον αφορά τις ασφαλίσεις. Και δεν θέλουμε να μαντεύσουμε ποια θα είναι η απάντηση. Θα δούμε τι γίνεται συγκεκριμένα με τις ασφαλίσεις αφού ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά τις υποχρεώσεις και μετά θα δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού. Πολύ δουλειά ακόμα θα τελειώσει το 2010-2011 η δουλειά, δεν θα τελειώσει μέχρι το τέλος ε, τρέχοντος έτους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πάμε σε ένα-δύο ε, ερωτήσεις από την ομάδα σοσιαλιστών. Ο κύριος Σάνσες Πεσάδο. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ ότι είσαστε παρόν εδώ. Ουσιαστικά οι πτυχές οι είναι ένα από τα κέρια θέματα όταν εξετάζουμε αυτή την κρίση την οικονομική. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να γίνει κάποια αναφορά για την ε, εξέλιξη της διαχείρισης την εξέλιξη των θεμάτων διαχείρισης. Μια και τόσο η Ευρωβουλή όπως και η Λέσχη των 20 στην συνάντησή τους ε, έχουν θέσει τα διάφορα σενάρια για τους holders. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται σε σχέση με αυτή την πτυχή και ταυτόχρονα για τη συμφωνία που επετεύχθη για την χρηματοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μια προοπτική από πλευρά μια αναφορά σχετικά. Επίσης είναι σημαντικό, πιστεύουμε, το επίπεδο όπου αυτές οι προδιαγραφές θα υιοθετηθούν από τρίτες χώρες. Θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά επίσης και σε αυτό το θέμα. Και όσον αφορά επίσης τη συνεργασία, συνεργασία με τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό είναι κέρια σημασία, θεμελιώδου σημασία για να υπάρξει ένα διεθνέ λογιστικό σύστημα επιτήρηση. Θα ήθελα να μου πείτε από τι επαφέ που είχατε μέχρι σήμερα, υπάρχουν κάποιε διαφορέ ω προ αυτά τα θέματα. Και ποιε θα ήταν οι πιο διαφορετικέ, θα έλεγα, εναλλακτικέ λύσει. Και υπάρχει μια δυνατότητα συμβιβασμού, συμφιλίωση μεταξύ των διαφορετικών σεναρίων. Και θα ήθελα επίση, αν γίνεται, να μου αναφέρετε να κάνετε κάποια αναφορά για το ποιο είναι το πρόγραμμα της άμεσης προσαρμογής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε. Καυτά τα θέματα που θίξατε. Τα πρώτα δύο ζητήματα είναι θέματα των διαπιστευτών. Παραδιακυβέρνηση πρέπει να δείτε τι γίνεται με το θεσμό μας. Όταν δημιουργηθήκαμε, οι βασικοί φορείς που σχημάτισαν το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το SEC και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό το Συμβούλιο, το Διοικητικό, βασίστηκε στα πρότυπα των Αμερικανών, με μια μεγάλη διαφορά όμως. Είχαμε ανεξάρτητο Συμβούλιο που έπαιρνε αποφάσεις διάφορους μετόχους που δεν μπορούσαν να σε τεχνικά θέματα και διόριζαν τους διαδόχους τους. Αυτό που έλειπε ήταν αυτό που είχαν οι Αμερικανοί, το SEC δηλαδή, ο φορέας που διοριζόταν από τα δημοκρατικώς εκλεγμένα μέλη. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο να γίνει για διεθνή φορέα, διότι δεν υπήρχε το διεθνές SCC. Και σε αυτή τη φάση ελάχιστες χώρες χρησιμοποιούσαν αυτά τα πρότυπα. Ήταν βήμα προόδου πράγματι το ότι πέρσι δημιουργήθηκε το, συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο Εκεί εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και με τους ρυθμιστές των, τους, Ιαπών, τους Ιάπωνες, τον πρόεδρο των SEC και άλλους ανώτερους επόπτες, εποπτικούς φορείς από την ΕΟΣΚΟ. Η Βασιλεία συμμετέχει ως παρατηρητής. αυτή ήταν, αυτό ήταν το αρχικό σχήμα, αλλά θα συζητηθεί ε, αλλά τώρα έχουμε κάπως διασυνδεθεί με τη δημοκρατική διαδικασία κάτι που απασχολούσε αυτή την Επιτροπή και αυτό έπρεπε πράγματι να συμβεί. Ήταν σωστό και δίκαιο. Τώρα αν είναι σωστή η μορφή, αν είναι δεδειγμένη η μορφή, αυτό είναι θέμα προσυζήτηση. Χρηματοδότηση, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Κοστίζουμε περίπου 15-18 εκατομμύρια λίρες το χρόνο για λειτουργικά έξοδα. Και έχουμε έλλειμμα δεν έχουμε αρκετή χρηματοδότηση, διότι η χρηματοδότηση δεν έρχεται από τη ΣΥΠΑ. Εν φταίει αυτό, αλλά και από την Ευρώπη ακόμα. Δεν είναι πολύ γενναιόδορη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα δώσει κάποια χρήματα του χρόνου, αλλά λιγότερα από αυτά που παίρνουμε από τι διάφορε χώρε για την ώρα. Αυτό είναι κάτι που μα προβληματίζει και σίγουρα θα θέλουν να μα μιλήσουν για το θέμα αυτό. Η χρηματοδότηση λοιπόν είναι κάτι που μα προβληματίζει. Συνεργαζόμαστε με άλλου διεθνεί φορεί Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει λοιπόν με το κόστος. Έχουμε πρόβλημα χρηματοδοτικό. Άλλες χώρες, προανέφερα τις διάφορες χώρες που συμμετέχουν. Αν δείτε ένα χάρτη παγκόσμιο, θα δείτε ότι η Λατινική Αμερική ε, μπαίνει όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η Ασία είναι ισχυρότατη, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη στην Ασία. Δημιούργησαν μια ομάδα που θα συζητά θα γίνεται συζήτηση των μελών. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος τη Ασία, δεν είναι οργανωμένοι το τρόπο, αλλά θέλουν να συζητήσουν μαζί μας. Και τρίτο κομμάτι είναι η ΕΠΑ. Και αυτό είναι το άλλο θέμα που θίξατε. Την περασμένη εβδομάδα η SEC, ο πρόεδρος της ΕΣΥ και ο αρχιλογιστής σχολίασαν και είπαν ότι ο δικό χάρτης της προηγούμενη κυβερνήσεω για να κινηθούν οι ΙΠΑ προς συμμόρφωση με διεθνεί προδιαγραφέ. δεν ήταν κάτι νεκρό ότι το φθινόπωρο θα προβούν σε σχετική δήλωση όσον αφορά αυτή την πρόταση και υποψιάζομαι ότι θα παραμείνει ζωντανό ο δικό χάρτης δεν έχω άλλες πληροφορίες επεξεργαζόμαστε πρόγραμμα σύγκληση που υπογράψαμε είπα και εμείς και θέλουν οι G20 να διεκπαιρώσουν τις εργασίε μέχρι το 2011 και ο δικός χάρτης προβλέπει ότι το 2011 θα ληφθεί απόφαση κατά πόσο οι ΕΠΑ θα πάνε στα IFRS και αυτό είναι το βασικό θέμα. Εάν δεν αλλάξουν οι ΕΠΑ τότε η συνεργασία με τι ΗΠΑ θα μειωθεί διότι ο υπόλοιπο κόσμος δεν θα ανεχθεί μια χώρα να εξοικονομεί πολύ χρήματα διότι δεν συμμετέχει. Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θα εξετάσουν τα θέματα, θα προχωρήσουμε προς τις προδιαγραφές, θέλουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα εργασιών, εμείς και δεν έχουν λόγο εκείνοι να μην ολοκληρώσουν. Άμα τελειώσουμε εμείς, τα αμερικανικά πρότυπα και τα δικά μας πρότυπα θα οδηγούν σε παρόμοια απάντηση. Έχουν 17.000 σελίδε πρότυπα. Εμεί έχουμε 2.500 σελίδε. Δεν είναι ακριβώ για τα πράγματα. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε στι 17.000 σελίδε με πρότυπα. Αλλά αυτό είναι το βασικό. Θα είναι ευκολότερο για αυτούς να κινηθούν αφού πάρουν σχετική απόφαση και εγώ ελπίζω ότι το 2011 θα πάρουν την απόφαση. Οι Ιαπώνες επιτρέπουν σε Ιαπωνικές εταιρείες να χρησιμοποιούν διεθνείς προδιαγραφές από φέτο και θα λάβουν τελική απόφαση για αλλαγή το 2012. Αλλά η απόφαση σχεδόν έχει ληφθεί, διότι πιο σημαντικές εταιρείε ήδη αλλάζουν ή ετοιμάζονται για να κάνουν την ε, αλλαγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κάθριν Στήλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ Σερ Ντέιβιντ για τις διεξοδικότατες απαντήσεις σας. Έχω κάποιες σύντομες ερωτήσεις. Μία από αυτές την αναφέρατε, το θέμα της συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ και το χρονοδιάγραμμα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε σαν Επιτροπή και σαν μέλη, διότι είμαστε και στην αντιπροσωπεία για τη ΣΥΠΑ, για να ασκήσουμε πίεση, ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα είναι κάτι χρήσιμο. Αυτό είναι πρακτικό μέτρο που μπορεί να ληφθεί. Πρώτα απ' όλα, έχω ερώτηση. Τι γίνεται με τις τράπεζες ε, η Lehman Brothers, ε, η ρευστοποίηση τη Lehman Brothers θα χρειαστεί μια δεκαετία. Δεν ξέρουμε ακόμα πού είναι τα χρήματα. Ποια είναι η υποψή σα, για το hedging. Είπατε τέλο του χρόνου θα υπάρξουν απόψει και θα είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα διότι θα υποβληθούν και προτάσει από την Επιτροπή για διάφορα νομοθετήματα σχετικά με αυτό. Και αυτά που είπατε και για τι ασφαλιστικέ εταιρείε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τι θέλουμε εμεί. Πολλοί από εμά στην Επιτροπή συζητούμε παγκόσμιε προδιαγραφέ και πρότυπα και σίγουρα δημιουργείται ένα προηγούμενο πάνω σε αυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να σα βοηθήσουμε σε αυτό είναι χρήσιμο. Και τέλο, όταν επιστρέψετε τι Ευρύδε, εγώ εκπροσωπώ τη Σκοτία, να δείτε πώς δουλεύει το ευρυζωνικό εκεί πέρα. Διότι μπορείτε να δείτε τι μπορεί να γίνει με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στι Ευρύδε για το θέμα των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αναγνώρισα την προφορά σας πριν μου είπατε από πού κατάγεστε. Κοιτάξτε, η κατάσταση για τη Lehman Brothers Όλοι μάθαμε μάθημα αυτό. Ξέρω ότι το Συμβούλιο για την Οικονομική Σταθερότητα το συζήτησε το θέμα, για την σταθερότητα και κυβερνήσει όλο τον κόσμο απασχολούνται για το πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Πόσο περίπλοκοι είναι αυτή η φορεί. Και γίνεται προσπάθεια για να αφαιρεθεί αυτό ο περίπλοκο χαρακτήρα, οι θηγατρικέ, τα holdings και όλα αυτά, να είναι απλούστερε οι δομέ. Οπότε αυτό θα ισχύσει σε όλη τη χρηματοπιστωτική κοινότητα. Και για τα παράγωγα, τα μέσα των παραγόγων ήταν πάρα πολύ περίπλοκα και ο κόσμο δεν τα καταλάβαινε. Και φαντάζομαι ότι η αγορά θα μειωθεί για αυτά τα προϊόντα. Δεν τα αγοράζει ο κόσμο έχοντα δει τι συνέβη. Άρα γίνονται προσπάθειε όχι από εμά αλλά από άλλου που προσπαθούν να εξετάσουν αυτό το τομέα. Τώρα το θέμα του hedging είναι ένα κομμάτι των λογιστικών που είναι περιπλοκότατο και δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο. Υπάρχουν δύο διαφορετικέ μέθοδοι για το hedging. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία μέθοδο και μόνο. Δεύτερον, έχουμε δοκιμή αποτελεσματικότητα να χρησιμοποιήσει λογιστικά hedging, δηλαδή να αναβάλει τον υπολογισμό κερδών και απολύων για επόμενα έτη, για να λάβει υπόψη το hedging. Αν λοιπόν το hedging σου είναι αποτελεσματικό λιγότερο από 80% δεν μπορεί να προστατεύσει, δεν μπορεί να κάνει hedging. Αυτό είναι ένα κανόνα. Γιατί είμαστε 70% αποτελεσματικότητα, 70% 60%. Αυτό εξετάζουμε, προσπαθούμε να μειώσουμε την περιπλοκότητα του ζητήματος και ελπίζουμε να μας δοθούν περίπου αρχέ του επόμενου έτου κάποιε απαντήσει. Αυτό είναι που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αργότερα αν επιθυμείτε. Ελπίζουμε λοιπόν ότι πάντως... Και το, η δική μου ευρυζωνική σύνδεση δεν δουλεύει καλά και είμαι κοντά στο Εδιμβούργο. Έχω και εγώ πρόβλημα. Η Βίκη Φόρντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Σερ David. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να διαβάσει κανείς σήμερα το Financial Times γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο λέγεται ότι ε, δεν πιστεύει κανείς πλέον τις τράπεζες και δεν νομίζω ότι αξίζει να είναι επικεφαλίδα μιας εφημερίδας αλλά γι' αυτό εσείς ε, σαν λογιστές πρέπει να βοηθήσετε και να διευκρινίσετε την ανάγνωση των ισολογισμών. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνέπεια, σαφήνεια ε, και βεβαιότητα διότι με ανησυχία ανησυχεί πάρα πολύ ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση ε, για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα λογιστικά πρότυπα στην Αμερική και στην Ευρώπη και ε, θα ήθελα να ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε για να ακολουθήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Στο παρελθόν, πριν από χρόνια, δεν είναι η παρούσα μου δραστηριότητα, είχα ε, ασχοληθεί με τις αγορές που έχουν μη ρευστοποιήσει χρεόγραφα. Μία ε, ε, αγορά η οποία είναι πολύ ασαφής και πολύ αβέβαιη. Οπότε νομίζω ότι ανησύχησα, ε, μπορείτε να καταλάβετε ότι ανησύχησα ότι υπάρχουν πολλά περιουσιακά στοιχεία τα οποία μετατίθενται εις χώρες όπου τα λογιστικά πρότυπα υπολογίζουν το κόστος κτίσεως των ε, περιουσιακών στοιχείων και ότι εάν ε, ε, δημιουργηθούν χρεόγραφα χρησιμοποιούνται όμο χρησιμοποιούν μία μορφή η οποία βασίζεται εις το κόστος της αγοράς θα ήθελα λοιπόν να ξέρω επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι πολιτικά και οικονομικά δεν πρέπει να αναστραφούν αυτά τα οποία έχουν γίνει θα ήθελα λοιπόν να ξέρω γιατί αναστράφησαν αυτά που είχαν γίνει πέρυσι και τι επιπτώσεις οικονομικές μπορούν να έχουν. Ευχαριστώ όσον αφορά την περιπλοκή. Τα λογιστικά δεν είναι μια θετική επιστήμη και αν διαβάσετε τα διάφορα έγγραφα αυτά έχετε τέσσερις κατηγορίες που δεν χρειάζεστε. Έχουμε διαφορές με τις Ηνωμένε Πολιτείε οι οποίες προτείνουν τώρα να υπάρχει η σωστή αξία σε όλα τα χρεόγραφα και έχουμε, πρόκειται να έχουμε σε ένα μήνα μία συνάντηση όπου θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα θέματα. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν δύο κατηγορίες, μία υπολογισμός βάση του κόστους και μία βάση της αποτιμήσεως της σωστής αξίας. Οπότε ε, θα, με την τωρινή πρόταση μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο δηλαδή μπορείτε να αποκαλύψετε περισσότερα στοιχεία να βρείτε αυτά τα οποία δίνουν και οι Αμερικάνοι αλλά όπως είπατε όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι πολύ σαφής η κατάσταση έχουμε 20 οργανώσεις και ρωτήσαμε τους ε, ε, ελεγκτές, του λογιστές τους ε, ε, ρυθμιστές οι οποίοι ε, έχουν ελέγξει τα βιβλία και βλέπουμε ότι ο καθένας καταλήγει σε διαφορετικά αποτέλεσμα παρόλο που προσπαθούν όλοι να κάνουν περίπου το ίδιο. Πιο επιτυχής είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα πρότυπο με την τιμή αγοράς αλλά όταν η αγορά στέρεψε είχαν προβλήματα και είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε διότι υπάρχει μεν ένα κέρδος, αλλά κέρδος από τι. Θέλετε να το αποτιμήσετε για το μέλλον, οπότε αντιλαμβανόμαστε το κίνδυνο. Ε, το κόστος δεν μας βοηθάει γιατί μπορεί να είναι δεσμευμένο και πάλι αυτό δεν μας βοηθάει. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό, άπαξ και έχουμε ε, απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Η securitization ε, την οποία αναφέρατε ε, προσπαθούμε να δούμε ε, ε, ε, τι στοιχεία κόστους είναι. Πρέπει ίσως πρέπει να ξεχωρίσουμε τα χλωρά από τα ξερά και για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Είναι επίσης κάτι το οποίο θα, θα κοιτάξουμε, οπότε μπορείτε να δείτε ε, εάν υπάρχει, υπάρχει κάτι τέτοιο.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 Παρακαλώ, ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Ε, για να αποκαταστήσουμε την, ε, την εμπιστοσύνη πρέπει να γίνουν διαφανείς η φορολογική παράδεση. Γνωρίζουμε ελάχιστα την νομοθεσία τους. Ορισμένοι τη χρησιμοποιούν για να μην πληρώσουν φόρο Νομίζω λοιπόν ότι είναι βασικό να τους υποχρεώσουμε να αναφέρουν κατά χώρα τα αποτελέσματα, τις δραστηριότητες και ε, τους ε, φόρους που κατεβλήθησαν. Διότι ε, είναι αδύνατον να μην μπορούμε να γνωρίζουμε τι πληρώνουν φόρους ε, οι εταιρείε στην Αγγόλα και στο Μαλί και ή ε, στο Λουξεμβούργο που υπάρχει η holding εταιρεία ε, για να μπορεί ο καθένας να γνωρίζει ε, τι καταβάλλεται στο δημόσια ταμεία. Θα ήθελα λοιπόν να δω και να μου πείτε εάν υπάρχουν πρότυπα τα οποία καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δυσκολίες και είναι βασικό για τις μεταφορές όταν γνωρίζουμε ότι 60% του διεθνούς εμπορίου περνάει ε, μεταξύ διαφόρων ομήλων και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να υπάρξει αυτή η διαφάνεια όντως είναι στην ημερήσια διάταξη και ε, συμφωνώ. Έγινε μία συζήτηση πριν από μερικά χρόνια, ίσως πέρυσι, και ελέγχθη ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε το, το πρόβλημα αυτό. Δεν υπήρχε το σωστό πρότυπο και γι' αυτό δεν συνενέσαμε. Αλλά στην ιστοσελίδα μας έχουμε διατυπώσει μία πρόταση για τις εξορυκτικές βιομηχανίες ε, για κάρβουνο, για πετρέλαιο κτλ. Ε, όπου ρωτούμε τι γίνεται με την ε, ε, κτήση ε, των φόρων από τις κυβερνήσεις διότι όπως ξέρετε ορισμένοι ε, γνωρίζουν και το ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα στην Αμερική υπάρχει μία, ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητάτε και εμείς θεωρούμε ότι στο σημείο αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα διότι υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν πολλοί λόγοι αλλά χρειαζόμαστε να συμφωνήσει η πολιτική, ε, η πολιτική δικαιοδοσία διότι διαφορετικά δεν θα κερδίσουμε τη μάχη. Εάν λοιπόν εσείς ε, θεωρείτε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καλό θα ήταν να μπορέσετε να βοηθηθείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, να, ε, να το επιτύχετε, διότι οι, Αμερικές η Αμερική μπορεί να το κάνει, αλλά ίσως θα έπρεπε και εμείς να το προωθήσουμε και θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και μια σαφής ερώτηση πολύ σύντομα. Μεταξύ των λίγων πραγμάτων που συμφώνησαν οι 20 είναι στο ότι πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο, να προοδεύσουμε στην έγκριση προδιαγραφών που θα, είναι, θα εγγυώνται την φερεγγιότητα των τραπεζών για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Αυτή η Ευρωβουλή πολύ σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσει την οδηγία απαιτήσεων κεφαλαίου Πράγμα που είναι δύσκολο, ε, δύσκολο να γίνει εφικτό αν δεν έχουμε σαφή λογιστικά πρότυπα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα που με ανησυχεί. Είναι το θέμα των ε, ε, κυκλικών εκείνων προβλέψεων ή στοιχείων που με διακριτική ευχέρεια αντιμετωπίζονται από πλευρά των εποπτικών αρχών των κρατών μελών σε σχέση με τους κινδύνους που αναφέρονται σε σχέση με δάνεια πιστώσεις. Χωρίς σαφή κριτήρια. Χωρίς σαφή κριτήρια είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε το τι γίνεται σε σχέση με τους επενδυτές, ιδιαίτερα με τους αλλοδαπούς επενδυτές υπάρχει έργο που γίνεται σε σχέση με, αυτές τις κυκλικές, ε, ε, με αυτά τα κυκλικά στοιχεία ώστε να υπάρξουν αντικειμενικές προβλέψεις και στοιχεία για ε, τις προβλέψεις και σε σχέση με τους κινδύνους που εμπλέκονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που το ρωτήσατε, διότι επεξεργαζόμαστε αυτό, εργαζόμαστε άκνος σε αυτή τη φάση. Θέλω να πω, συνδέεται και με τη δήλωσή μου. Κάναμε διάφορες κινήσεις κατά διάρκεια της κρίσης και αυτή είναι μία από αυτές. Παραδοσιακά η λογιστική χρησιμοποιεί συγκεκριμένο μοντέλο για τις απώλειες. Τις απώλειες που σημειώθηκαν. Δηλαδή όταν έχει ενδείξει ότι θα σημειωθούν απώλειες, προσπαθεί να τι καλύψει. Τι σημαίνει αυτό. Όχι όταν υπάρχει χρεοκοπία, αλλά υπάρχουν υπόνοιες για επερχόμενη χρεοκοπία. Ας πούμε υπάρχει μια κάμψη στην ε, παραγωγή πετρελαίου και υπάρχει μια πόλη που εξαρτάται στο Χιούστον, στο Αμπερντίν, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρεις ότι υπάρχουν απολύσεις. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν στεγαστικά δάνεια, θα μπορούν να πληρώσουν κλπ. Προσπαθεί να το καλύψει διότι τα στατιστικά στοιχεία στο λένε. Ακόμα και έτσι πιστεύουμε ότι ό,τι έγινε έγινε αργά. Συνέβη κρίση. Και όσο χειροτέρευαν τα πράγματα, ερχόταν και οι προβλέψεις που επιδίνουν την κατάσταση. Αν δει κανεί οι τράπεζε τώρα, Πώ τιμολογούν τα δάνεια. Αν θέλεις μια επιστροφή 7% και προβλέπεις απόλυση 2% θα χρεώσεις όλους τα δάνειά σου 9%. Προσπαθήσαμε με τις ρυθμιστικές αρχές να κάνουμε κάτι. Αν είχαμε ένα μοντέλο για αναμενόμενες απόλυες σε κάποια βάση, δηλαδή βάση εμπειρίας όσον αφορά το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, αναμένεις απόλυες 2%. Αντί τις καλές χρονιές να δείχνεις ότι έχεις 9% και ξαφνικά όταν σε χτυπάνε οι απώλειες δείχνεις 5-4-3, δεν θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσεις λέγοντας ξέρουμε ότι θα έχουμε τις απώλειες αυτές το πρώτο έτος στην τιμή θέλεις έσοδα 9% αλλά και 2% κάλυψη για τις επερχόμενες ε, απώλειες. Και μπαίνει και μέσα στο δάνειο, κατά τη διάρκεια του δάνειου, όχι στο τέλος την ε, τελική πληρωμή. Ε, κάναμε προτάσεις τον Ιούλιο, ζητήσαμε κάποια σχόλια, θα αλλάξουν πολλά συστήματα για να γίνουν αυτά που θέλουμε. Το συζητούμε αυτό, πώς θα πρέπει να γίνει. Οι αριθμιστικές αρχές πρέπει να μας βοηθήσουν. Είναι σωστό το 2%, 3%, 1%. Ποιο είναι το σωστό. Άρα θα είναι μια συζήτηση θα γίνει με τις ρυθμιστικές αρχές. Αλλά κινούμαστε σε αυτό το τομέα. Καλώς λέει η πρόεδρος. Επόμενος. Εγώ. Πάμε πίσω. Στο θέμα του fair value. όλα ακούγονται ότι είναι ελεγχόμενα όπως μας τα εξηγείτε. Αλλά είναι επίμαχος μάλλον και θα παραμείνει επίμαχος αυτός ο τομέας. Και ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το fair value όλο και περισσότερο, ώστε οι επενδυτές να γνωρίζουν πλήρως ποια είναι η αξία των επενδύσεών τους αλλά οι ρυθμιστικές αρχές για τη συνετή διαχείριση έχουν αρπάξει κατά κάποιο τρόπο τα πρότυπα αυτά τα λογιστικά, τα έχουν ενστερνιστεί, τα έχουν πάρει και υπάρχει μια ανάγκη να, για λόγους συνετής διαχείρισης να ληφθούν υπόψη με διαφορετικό τρόπο αυτά. Μήπως με συμβιβασμούς ενδιάμεσους θα λυθεί το πρόβλημα ή τελικά θα χρειαστεί να πούμε ότι για κάποια πράγματα θα πρέπει να προετοιμαστούμε ξεχωριστά άλλοι λογιστικοί υπολογισμοί για τους επενδυτές με διαφάνεια και μετά κάποιο συντελεστή μέσω XPRL λοιπά θα εφαρμόσουμε για να δούμε πώς θα υπάρξει αντιμετώπιση μέσω των κανόνων για συνετή διαχείριση και θα πρέπει να υπάρχει πανταχού διαφάνεια όλοι να ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Τι σκέφτεστε γι' αυτό. Δεύτερον, Αναφέρατε ακροφυγώς κάτι. Τα παράγωγα. Και τα OTCs και πώς ενδεχομένως τα αριθμιστούν. Έχετε κάποια λύση συγκεκριμένη. Με το νόμιμο hedging για τα παράγωγα μέσω των μεγάλων επιχειρήσεων, πώς κινήθηκαν. Ενδιαφέρονται πολύ για τα αξιόγραφα και κινούνται χωρίς να έχουν κερδοσκοπικό ε, σκοπό. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα. Πέστε μου αν το λύσατε. Απαντάω το τελευταίο. Δεν το λύσαμε. Το εξετάζουμε το θέμα. Και ελπίζουμε ότι στο τέλος του έτους, αρχές του επομένου έτους, κάτι θα δώσουμε πάνω σε αυτό σαν πρόταση. Όσον αφορά το θέμα συνετής διαχείρισης, κάτι που συνεκλώνησε τους περισσότερους όσον αφορά την κρίση, ήταν ότι τις καλές εποχές οι τράπεζες μοίραζαν τα κέρδη. Βόρεια Αμερική, Ευρώπη. Πώς το έκαναν. Μέσω ομολόγων, μέσω εξαγορών, μέσω αντισταθμίσεων. Άρα κράτησαν ελάχιστα κέρδη και γι' αυτό υπήρχαν μεγάλες πίεσεις. Πέρα από τις προσδοκόμενες απώλειες είπαν γιατί τον καιρό των παχιών αγελάδων δεν ε, ζητάτε μια εισφορά για τις ισχνές αγελάδες και χρησιμοποιείτε αυτά τα χρήματα. Πρέπει να καταλάβετε τι ζητούμε. Δηλαδή, χάνουν οι τράπεζες σε κακές εποχές και δεν είναι καλό για τις αγορές αυτό. Καταλαβαίνουμε τι προσπαθούν να κάνουν οι αρχές. Και μπορούμε και οι δύο να κερδίσουμε. Πώς? Να πούμε από τα κέρδη, χ της 100 δεν είναι διαθέσιμο για ανακατανομή ή αμοιβή μπορεί να είναι ελαστικό κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιείται σε κακές στιγμές μαζί με τη Βασιλεία. Και κάτι άλλο που αναφέραμε για το μοντέλο Fair Value έχουν φαίνεται διανεμηθεί και αυτά τα κέρδη. Μπορώ να το εξετάσουμε. Και τι γίνεται με τα έσοδα. Παίρνεις το κέρδος και λες ναι μεν, αλλά φερούμε ένα ποσό για κατανομή και αποζημίωση που μπορεί αυτό να αποτελείται από ό,τι αφήνει στην άκρη για κακές εποχές και για τη διαμόρφωση του μοντέλου. Χρειάζεται ρυθμιστικό εισόδημα μαζί με το επενδυτικό εισόδημα, αν θέλετε, δύο ειδών εισοδήματα. Δηλαδή γίνεται ένα είδος διχάλας, μπορείτε να το αποκαλέσουμε έτσι, ψαλίδα. Δύο αγορητές έχω στον κατάλογο και μας τελειώνει και ο χρόνος και παρακαλώ ακούσουμε και τους δύο πριν ο Σερ Ντέιβιντ δώσει απαντήσεις. Τζέφρι Μπλουμ πρώτο. και ο Λεωνάρντο Δημήτρη μετά. μετά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε Σερ Ντέιβιντ. Θα με ενδιαφέρει η παρατήρησή σα σε σχέση με περισσότερο από τη σε μια ερώτηση όσον αφορά τι διεθνεί ε, λογιστικέ προδιαγραφέ. Θα έπρεπε επίση να στραφούμε προς τις κυβερνήσεις για να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται οι σωστές αυτές λογιστικές αρχές. Δεν μπορώ να ομιλήσω εξ ονόματος άλλων. Ίσως μία αναφορά στη ΣΥΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να γίνει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, αναέτος είχαμε στοιχεία τα οποία δημιουργούσαν προβλήματα ιδιαίτερα όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, τον δανεισμό δημόσιου τομέα και θα πρότεινα σε, μια και ό,τι είναι ε, καλό για τον έναν είναι καλό για τον άλλον, πρέπει αυτό να επιβάλλεται με τον ορθό τρόπο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Μια διευκρίνηση θα ήθελα από πλευρά του Σερ David Tweety. Αν κατάλαβα καλά, η μεταρρύθμιση της αρχής των λογιστικών υπολογισμών θα έχει διάφορε στάδια που θα περάσει βήματα. Για ταξινόμηση, εξολόγηση των χρηματοπιστωτικών μέσων, για τον υπολογισμό τη απώλεια αξιών και για τι προσπάθειε κάλυψη. Το πρόβλημα είναι ποιο συντονισμό χρονικά υπάρχει. Μέχρι το 2012 θα καταβληθεί αυτή η προσπάθεια, αν κατάλαβα. Το, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι σε θέση να δώσει εγγυήσει ούτω ώστε να μην εντοπιστούν ξεχωριστά οι διάφορες πτυχές της αναθεώρησης των λογιστικών ε, υπολογισμών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των αλλαγών στο OEIS 39 θα πρέπει να έχει δυνητική ισχύ, εθελοντικά θα πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό ίσως θα χρειαζόταν να προβλεφθεί μια περίοδος εντός της οποίας θα συνεπάρχουν οι παλιοί κανόνες και οι νέοι κανόνες και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα για τους φορείς εκείνους για τους οποίους η εξή των προϋπολογισμών δεν στρέφεται γύρω από την αγορά και μόνο, αλλά και υπάρχει και θέμα νομικής αξίας για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, του φορολογούμενου εισοδήματος και των φορολογικών εσόδων. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα Τελευταία ερώτηση πρώτα διότι εδώ ήταν και το θέμα των λογιστικών προδιαγραφών όσον αφορά τις ε, καταγραφές ε, της κυβέρνησης ε, και αυτό ήταν σαν χειροβομβίδα. Αν μπορεί κανείς να δει τα, τον πίνακα για το 2012 για τα παράγωγα, δεν θέλησαμε να έχουμε μια πρώιμη, αν θέλετε, πρόβλεψη γιατί θα μπορούσαν να υπάρξουν στρεβλώσεις μπορεί αυτό το 2013 να γίνει, διότι πολλές χώρες το 2011 θα αλλάξουν ε, προς ε, ένα νέο πρότυπο και δεν θα πρέπει διαμιάς να γίνει αυτό, αλλά ε, σταδιακά. Και θα το δούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με διαφορετικούς κανόνες που συνεπάρχουν και γι' αυτό θα πρέπει να είναι σαφείς οι προδιαγραφές που θα ισχύουν. Και μπορεί να υπάρχει και διαφορετική αρχή που θα πρέπει να αποφασίζει το τι θα συμβαίνει σε διαφορετικές καταστάσεις και πότε κάποιες επιχειρήσεις μπορούν ή όχι να χρησιμοποιούν κάποιες τέτοιες προδιαγραφές. Θα ε, είναι δυνατόν σε κάποια διαχωριστική γραμμή να, να τεθεί κάποια διαχωριστική γραμμή χρονικά για το ποια πρότυπα θα ε, υιοθετούνται. Και νομίζω ότι αυτό είναι θέμα της Ευρώπης και αυτή τη δική σα κοινοβουλευτικής επιτροπής να υποβάλει συστάσεις. Αλλά για οποιαδήποτε θέματα αλλαγών όταν πρόκειται αυτές να γίνουν θα ληφθούν αυτά υπόψη. Όσον αφορά τις κυβερνήσεις τώρα όταν εξετάζει κανείς ε, τα λογιστικά σε σχέση με τις ε, κυβερνητικές καταχωρήσεις ε, υπάρχει τάση να διασφαλίζεται ότι και ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας θα υιοθετεί τα, τις ίδιες προδιαγραφές και για την Επιτροπή των Λογιστικών σε σχέση με την, την καταχώρηση λογιστικών προδιαγραφών του δημόσιου και υπάρχει επιχείρημα να χρησιμοποιούνται κοινέ προδιαγραφές για όλες τις καταχωρήσεις. Αυτό τώρα δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο όταν ε, είχαμε το θέμα των λογιστικών καταγραφών ε, των συντάξεων ε, και όταν υπήρχαν ελλείψεις και δημιουργήθηκαν επικρίσεις όταν όμως είχαμε μετά από κάποια χρόνια από ανώτερους υπαλλήλους ότι την παρατήρηση ότι επιτέλους συζητούνται κάποια θέματα αυτό για να σας δείξω τι μπορεί να συμβεί αν δεν είναι σωστές οι προδιαγραφές σας στα λογιστικά να δει κανείς την General Motors παρήχαν υγειονομική περίθαλψη στους εργαζομένους ε, σε σχέση με την συνταξιοδότησή τους. Ε, είναι πάρα πολύ δαπανηρό το θέμα της ε, υγειονομικής ασφάλισης και αυτό ήταν με το Pay As You Go Scheme. Και υπήρξε η παρατήρηση ότι εφόσον υπάρχει συνταξιοδότηση πρέπει να αναφέρεται η επιβάρυνση αυτή. 32 δις δολάρια και αυτό είναι τεράστιο ποσό και γίνεται λόγος επίσης για το ότι για κάθε αυτοκίνητο της General Motors που πωλείται τεράστιο ποσό παρακρατείται για, τους, για τις συντάξεις των συνταξιοδοτημένων εργαζομένων. Και είναι αυτό δυσανάλογο ποσό σε σχέση για παράδειγμα με την Ιαπωνία. Αυτό πρέπει να δούμε ως πρόβλημα και να το, με τις καταχωρήσεις συλλογιστικές να επιλυθεί. Φυσικά τώρα θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα σε σχέση με τις λογιστικές καταγραφές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι να μην υπάρχει αποκάλυψη και να μην υπάρχει αποσιώπηση. Πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια αυτό. Και σε σχέση με τα ελλείμματα όσον αφορά την κάλυψη, τη συνταξιδοτική και την υγειονομική, πρέπει να αυτά να αποκαλύπτονται. Σας ευχαριστώ, Σερ Ντέιβιτ. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντική η παρουσία σας και μπορέσαμε μέσα στο, ε, χρόνο που είχαμε σε μια ώρα να ε, καλύψουμε τις ανάγκες μας. Θα λάβουμε υπόψη την προσφορά σας να, επανέλθετε στην Κοινοβουλευτική μας ε, Επιτροπή και να έχουμε την δυνατότητα μέσω σεμιναρίου ή οποιασδήποτε τέτοια επαφή να ανανεώσουμε αυτές τις συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στο επανειδή. Χάσαμε κάποιο χρόνο, καθυστερήσαμε λίγο και τώρα πρέπει, έχουμε ένα τέταρτο ακόμα, προτού έρθει ο κύριος Τρισέ στη συνεδρίασή μας. Σημείο 6 στην ημερησία διάταξη είναι οι δυνατότητες μικροδανείων και χρηματοδότησης για την κοινωνική ένταξη. Εισηγητής ο κύριος Όλε Σμιτ Νομίζω είναι έτοιμος να παρουσιάσει την έκθεσή του. Έτσι του δίνω τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσοι από εσά είσαστε εδώ παρόντε στο παρελθόν, γνωρίζετε ότι είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και στο παρελθόν στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή. Ο πρώην συνάδελφο Μπάξη είχε ασχοληθεί με μια έκθεση για τα μικροδάνεια, μικροπιστώσει. Υπάρχουν και άλλα έντυπα, έγγραφα και πρωτοβουλίε και πριν από αυτό. Και τώρα υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση, μια απόφαση. Είναι μια γνωμοδότηση. Η ε, επί της ουσίας αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή είναι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η δική μου πρόταση ποια είναι. Λέω να δεχθούμε αυτή την πρόταση της Επιτροπής και να συμφωνήσουμε κυρίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αδρές γραμμές. Είναι, μπορεί να είναι ένα ευαίσθητο θέμα και αν θέλουμε να ασκήσουμε κάποια επιρροή και να γίνει κάτι πρέπει γοργά να δράσουμε σε αυτό το επίπεδο και να μην χρονοβορήσουμε και περιμένουμε και καθυστερούμε. Πρότασή μου είναι να δεχθούμε λοιπόν την πρόταση της Επιτροπής. Γνωρίζουμε ότι οι μικροπιστώσεις τα μικροδάνεια έχουν θεμελιώδη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις και ξέρουμε ότι τέτοιου είδους μικρές επιχειρήσεις έχουν δεσπόζοντα ρόλο στην Ευρώπη. Υπάρχει ένας ορισμός που μπορούμε να δεχθούμε και τον δεχτήκαμε και την τελευταία φορά μικρότερες από 25.000 ε, ευρώ και με λιγότερους από 10 ε, εργαζόμενους και πρέπει έτσι στοχοθετημένα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο να ασχοληθούμε και σε σχέση με τους μη απασχολούμενους, τους άνεργους που θέλουν να μπορέσουν να αυτοαπασχοληθούν και πρέπει να βρούμε χωρίς ε, γραφειοκρατική επιβάρυνση τρόπους και δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ίσως κάποια προβλήματα, όμως ε, ε, φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι φορείς σε επαφές και συζητήσεις, αυτοί οι φορείς θα πρέπει να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και να παράσχουν ένα πλαίσιο στήριξης ώστε αυτού του είδους οι ε, πιστώσεις, ε, τα δάνεια στα 27 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζονται. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ε, μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και πρέπει όλα να γίνουν γοργά. Ίσως κάποια άλλα θέματα σε σχέση με την Ευρωβουλή οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θέλουν ένα νέο κονδύλιο στον προϋπολογισμό. Θέλουν επιπρόσθετα κονδύλια να διασφαλιστούν γι' αυτό. Και από τουλάχιστον όσα έχω δει δεν θα δεχθούν αυτή την πρόταση που υποβάλλουμε. Η πρόταση σε εσά συνάδελφοι είναι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι θα πρέπει να δεχθούμε αυτή την πρόταση. 100 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν ως κονδύλιο για μια τετραετή περίοδο. Και θα υπάρξει δυνατότητα και χρηματοδότηση ε, επιπρόσθετα και από άλλες πηγές. Αυτό το ειδικό ξεχωριστό πρόγραμμα, το πρόγραμμα του μέσου για τις μικροπιστώσεις και μικροδάνεια, ε, αφορά αυτό το ποσό. Κάποιες ε, μικρές αλλαγές στον ορισμό γίνονται, μπορούν να γίνουν και με μια άλλη τροπολογία, αλλά σε αδρές γραμμές μπορώ να πω ότι υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία. προβληματίστηκα επιπλέον και για μηχανισμό ελέγχου και δυνατότητες αντιμετώπισης απατών και διαφθοράς ή ε, στρεβλών πρακτικών να υπάρξει μια σωστή εποπτεία διότι πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χρήση αυτών των κονδυλίων των κονδυλίων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Φυσικά δεν είναι τεράστιο αυτό το ποσό. Μπορεί κανείς να συζητήσει για 100 εκατομμύρια ή για 150 εκατομμύρια ευρώ. <clears throat> Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε και τα 27 διαφορετικά κράτη-μέλη. Δεν είμαι απόλυτα πεισμένος ότι <clears throat> εξάλλου για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης δεν θα είναι αυτό η κύρια πρωτοβουλία αλλά είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και θα έπρεπε να το κάνουμε και γοργά αν γίνεται να μην καθυστερήσουμε θα ήταν ανόητο, θα έλεγα, να απορρίψουμε αυτή την πρόταση σήμερα, λέγοντας δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να τα δούμε και, ότι χρειάζεται μια ευρύτερη προοπτική αν κάναμε κάτι τέτοιο και το απορρίπταμε δεν θα βοηθούσαμε εκείνους που χρειάζονται την υποστήριξή μα, ε, και στο σύνολο τη Ευρώπη πρέπει να βοηθηθούν. Η κύρια ευθύνη φυσικά είναι των κρατών μελών και των διαφορετικών κυβερνήσεων των κρατών μελών και των συναδέλφων μα βουλευτών στα κοινοβούλια των 27 κρατών μελών τη Ένωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει θετικά να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα. Εμεί είμαστε εκείνοι κατά τα άλλα που υποστηρίζαμε και ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει μια πρωτοβουλία και να κάνει κάτι. Και η έκθεση μπάξη τον ε, Μάρτιο ε, εφέτος ε, ήταν ακριβώς κάτι που ήταν πρόταση της Ευρωβουλής σχετικά. Θα ήταν ανόητο λοιπόν να μην δεχόμαστε, να μην δεχθούμε την πρόταση αυτή σήμερα. Παρότι φυσικά μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές απόψεων. Εν συμπερασματικά διατάφτα. Με τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Ο κύριος Γκοζές. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θα ήθελα να μιλήσω για να ζητήσω συγγνώμη κυρία Ρόδη Κράτσα που είναι σκιώδη συγγήτρια για την ομάδα μας. Θα ήθελα να σας πω και σε εσάς και συναδέλφους αυτά που θα υποθούν σήμερα θα τις θα διαβιβάσω με πιστότητα για να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στην αποστολή της. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για αυτή την πρόταση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χώρα μου, η Λετωνία, είναι μια από τις χώρες εκείνες που επλήγησαν ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα της επιπτώσης οικονομικής κρίσης. Ε, είναι τεράστιος ο αριθμός. 90% ε, των λετωνών ε, υπηκών που εργάζονται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 απασχολούμενους. Οι, τα πιστοτικά ιδρύματα, οι τράπεζες δεν διαθέτουν, δεν δίνουν πια τέτοιου είδους δάνεια. Δεν είναι θέμα ποσοστών ή παράλληλης τέτοιας χρηματοδότησης, αλλά δεν μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να βοηθηθούν και να ξαναστηθούν στα πόδια τους. Και ένα μέσο, μέσο του προϋπολογισμού, εδώ έχουμε και ένα μικρό ποσό, 100 εκατομμύρια για τις, τα, τις μικροπιστώσεις, μικροδάνεια, έχει τεράστια σημασία. Δεν είναι μόνο για τη Λετωνία, σίγουρα για όλα τα κράτη-μέλη αυτό. Εντάξει, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων εργάζονται σε αυτές τις ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να τολίσω λοιπόν την σημασία της ταχύτητας. Γοργά να δράσουμε, ταχύτατα να υποστηρίξουμε όσους χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. το νόημα και ο στόχος αυτού του μέσου και η πρόταση της Ευρωπαϊκής είναι τα χρήματα αυτά να πάνε στις μικρές επιχειρήσεις όσο το δυνατόν πιο γοργά και έτσι η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει έντονα να υποστηρίξει αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, Σας ευχαριστώ. Περβάνος Σμπερέ στη συνέχεια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεώρησα ότι συνήθως δίναμε πρώτοι στους κοιόδης ηγητές το λόγο. είμαι σκιώδη συγγήτρια εκ μέσω σοσιαλιστών. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την ποιότητα της πρότασής του και θα ήθελα να καλέσω να προχωρήσει σαν δελεχέστερο προβληματισμό και να μας εξηγήσει ποια είναι, ποιο είναι το πνεύμα της ε, προτάσεις που βάλετε. Κύριε Ισηγητά, σωστά υπενθυμίσατε ότι με την έκθεση Backjay ζητήσαμε και υποστηρίξαμε, υποχηματολογήσαμε, ούτως ώστε η δυνατότητα μικροπιστώσεων να εφαρμόζεται. Το κάναμε σε αυτή την Επιτροπή, το κάναμε και στην Επιτροπή Προπολογισμών με ένα σχέδιο πιλωτικό, πρόγραμμα πιλωτικό που είχε τον ίδιο σκοπό. Όσον αφορά τη γενική προσέγγιση που εξετάζουμε, όσον αφορά το μέσο αυτό για τις μικροπιστώσεις, υπάρχει ένας κίνδυνος. Δηλαδή, να μην θεωρηθεί σαν συμπληρωματική διευκόλυνση αυτή που θα βοηθά τις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και εν αυτή τη ενία ε, παρατείνουμε κάπως τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όμως πιστεύω ότι το μέσο αυτό για τις μικροπιστώσεις ε, είναι κάτι ξεχωριστό. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Θέλουμε να βοηθήσουμε να ξαναμπούν στην αγορά εργασία οι άνθρωποι, να γίνει επανένταξη, να υποστηρίξουμε την επιχειρηματική εφευρητικότητα. Για αυτούς που συμμετέχουν σε μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση. Να βοηθήσουμε αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα χρηματοδότησης. Θέλουμε συμπληρωματική προσέγγιση εν συγκρίση με αυτό που προτείνατε. Μακριά από η ιδέα να αρνηθούμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένα τέτοιο σχέδιο που ζητούσαμε και φωνάζαμε γι' αυτό επί σειρά ετών. Το να δεχτούμε όμω ένα πρόγραμμα και να το δεχθούμε ανεφόρων ε, είναι κάτι που χρήζει διαπραγματεύσεων. Μεταξύ αποδεχτούμε ένα πρόγραμμα άνευ και μετά κάποιων όρων. Και γι' αυτό σα καλώ να μπούμε σε διαπραγματεύσει. Έχουμε λίγο χρόνο. Ε, επιγραμματικά μιλάω, θα ήθελα να σε πιστεί την προσοχή σε τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο αφορά το κονδύλι επί το οποίο θα ενταχθεί αυτό το μέσο. Επί τη γραμμή αυτή. Τα ρούχα κάνουν τον παπά βέβαια, αλλά τι να πω. Ε, το πρόγραμμα Progress πρέπει να δούμε, που είναι στον τομέα τη αντιμετώπιση του αποκλεισμού και τη παινία και είναι ένα από τα σπάνια προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, που πρικοδοτείται. Και κάποια κράτη-μέλη διστάζουν στο να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι πιστώσει, αυτό το κονδύλι, ενώ θα μπορούσαν να υποβληθούν πολλέ αιτήσει. Και το Συμβούλιο θέλοντας να διευκολύνει το του και θέλοντας να ικανοποιήσει τα αιτήματα χρηματοδοτώντας τη γραμμή Progress είπε υπάρχουν χρήματα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή, το κονδύλι του Progress και για μικροπιστώσεις. Είναι διαφορετικά πράγματα. Χρειαζόμαστε δύο κονδύλια. Και γι' αυτό θέλω να υπάρξουν δύο νέα κονδύλια, να δοθούν περισσότερα χρήματα από αυτά που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή μας μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια προσέγγιση. Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μάλιστα με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτόν τον σκοπό. Τέλος. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να καταπολεμηθεί η απάτη και η διαφθορά. 100% σας υποστηρίζω. Κοινό μας στόχος. Να πω και δύο άλλα πράγματα όμως που είναι κρίσιμη σημασίας. Πρώτα απ' όλα, η πρόσβαση στις μικροπιστώσεις. Πώς θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύει πώς διοργανώνουν τα κράτη-μέλη την πρόσβαση στις μικροπιστώσεις, διότι είναι κρίσιμη σημασία για τον προγραμματισμό και παρομοίως πώς θα συνοδεύονται εκείνοι που βρίσκονται σε πολύ εύθραστη κατάσταση. Πώς θα έχουν αυτή πρόσβαση στη χρηματοδότηση. πώ θα μπορούν να ανταποκρίνουν τις υποχρεώσει που αναλαμβάνουν. Αυτά κύριε Σιγητά. Θα προτείνω σχετικά κάποιες τροπολογίες και βάσει αυτών μπορούμε να καταλήξουμε ελπίζω σε κοινή θέση. Κοινή θέση ίσως ε, πιο που λαμβάνει, υποστήριξη, λαμβάνει υπόψη διάφορε λεπτομέρειε πέρα τη γενική υποστηρίξεω που προτείνεται. Ξέρω ότι να προχωρήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά στο Κοινοβούλιο χρειάζονται περισσότερε διαπραγματεύσει και με το Συμβούλιο πάνω απ' όλα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να βαθύνουμε στο θέμα. Έχω ένα πρόβλημα. Έχουμε τρία λεπτά και τρει ομιλητέ. Ο κύριο Μέντε Δεβίγο, κυρία Γεώργη και ο κύριο Μπαρόνε. Εστέ σύντομοι, παρακαλώ. Διαφορετικά θα πρέπει να σα διακόψω. Για να προλάβετε να μιλήσετε όλοι, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κοινοβουλευτική μα επιτροπή έχει τεράστια σημασία, αναφέρθηκε. Και ξεκινά τώρα η περικοπή χρόνου παρεμβάσεω σε ένα λεπτό και πρέπει να είναι πολύ ταλαντούχο κανεί για να μπορέσει να τα καταφέρει. Θα το δοκιμάσω, θα το προσπαθήσω, Πρόεδρε. Σε σχέση με την κυρία Μπερέ, ρώτησε ήδη κάτι που σε μένα δημιουργήθηκε αυτή η ερώτηση από την παρέμβαση του κυρίου Σμιτ. Γιατί η ανάγκη αυτής της ταχύτητα. και προηγούμενα αναφέρθηκε το θέμα ταχύτητα, Γιατί, δεύτερον, δεν μπορώ να κατανοήσω πάρα πολύ καλά γιατί υπάρχει αντίσταση σε ένα κονδύλι ε, προπολογισμού σαν αυτό να μου το αποσαφηνίσετε, γιατί δεν είναι απόλυτα σαφέ. και σε σχέση και με την παρέμβαση της κυρίας Μπερές επίσης. Και για αυτά που είπε ο κύριος Σμίτ, το 2010 το έτος για το, την καταπολέμηση της, του αποκλεισμού και τη στόχια, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί τέτοιου είδου ε, μέσα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινούνται το να κάνουμε δηλώσεις για έτη που θα αφιερώνουμε σε ένα συγκεκριμένο στόχο και μετά να μην ε, πρικοδοτούμε με μέσα και να μην δραστηριοποιούμαστε για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι δεν είναι το σωστότερο. Ένα λεπτό τήρησα, έκανα ό,τι μπορούσα. Καλύτερο, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Και εγώ έχω παρόμοια, στη χώρα μου έχουν παρόμοια προβλήματα όπως η Ετωνία. 88-94% των εταιριών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, άρα εκτίθενται πολύ σε κάθε κρίση που πλήττει τις εταιρείες τις πολύ μικρές. Θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα. Έλεγα λοιπόν... Συνεχίζει στα Ουγγρικά. Και θα ήθελα να ε, αναφέρω κάποιες σκέψεις. Όπως και ο κύριος Σμίτ, έτσι και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το μέσο θα πρέπει να πάρει τέτοια μορφή ώστε εκείνοι που έχουν χάσει τη θέση απασχόλησή τους να βοηθηθούν αλλά και εκείνοι που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και απειλούνται να χάσουν τη θέση απασχόλησης. Πρέπει τα διαθέσιμα κονδύλια να αναλωθούν στις ε, υφιστάμενες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, υπάρχουν διάφορες ε, δυνατότητες μικροδανείων στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή με 8,5% ποσοστό επιτοκίου. Είναι υπερβολικά υψηλό αυτό. Θα ήταν πολύ καλό αν θα ήταν δυνατόν τα ποσά που θα μεταφέρονται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με χαμηλά επιτόκια για τέτοιου είδους ε, μικροδάνεια. Τρίτον, υπάρχει και διαφορά απόψεων που υφίσταται μεταξύ μας σε σχέση με αυτά. Με την πρόταση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρόκειται να τα αναλάβει αυτά. Εμείς θα θέλαμε οι εθνικές τράπεζες ανάπτυξης να υπομισθούν αυτό το ρόλο, γιατί μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές. Και τέταρτον, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ε, ποιοι θα είναι οι κανονισμοί εφαρμογής, εκτελεστικοί κανονισμοί. Και σε σχέση με τα θέματα των, ε, που περιέπλεκαν τα πράγματα όσον αφορά αυτούς τους ε, κανόνες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην είμαστε υπερβολικοί όσον αφορά το γραφειοκρατικό βάρος που επιβάλλεται και να είναι ανέφικτη μετά η προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρόνε παρακαλώ εντάχει. Ναι, θα είμαι πραγματικά γρήγορος. Κάποιες σκέψεις ή κάποιοι προβληματισμοί είναι αυτοί που θέλω να κράσω κυρία Πρόεδρε όσον αφορά μια τροπολογία Σμιτ που προσπαθεί να διευρύνει το πεδίο των δικαιώχων και στις επιχειρήσεις που δεν έχουν κοινωνικό, κοινωνική επιρροή. Θα πρέπει να αποφύγουμε να αποδυναμώσουμε το θέμα. Θα πρέπει να καλύψουμε τις περιπτώσεις με άλλα μέσα υπάρχουν στις χώρες όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε τελείως την όλη ιδέα των μικροεπιχειρήσεων. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα διεθνή μέσα. Διεθνή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Παγκόσμια Τράπεζα επενδύσεων κλπ. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και πώς θα εφαρμόζεται και μέσω και των άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ε, το πρόβλημα αυτό των, μικρο... των μικροεπιχειρήσεων. Κύριε Σμιτ, θέλετε να απαντήσετε πάρα πολύ γρήγορα σε όλα αυτά που ετέθησαν. Ναι, άκουσα, σημείωσα όλα τα επιχειρήματα που ακούστηκαν Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις τροπολογίες και μετά βεβαίως ε, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση στο τέλος. Το πιο κρίσιμο είναι αυτό που είπε η πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης. Δηλαδή χρειάζεται περισσότερα χρήματα. Ίσως να είναι παρακινδυνευμένο αυτό. Θα δούμε όμως. Γι' αυτό δεν πρότεινα κάτι τέτοιο και γι' αυτό δεν πρότεινα κάποιο κονδύλι. Και αυτή ήταν η θέση του κυρίου Μπέκτσι τότε. Θα δούμε άμα καταφτάσουν οι τροπολογίες. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Είναι γνωμοδότηση αυτή. Γνωμοδότηση. Θα, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών η 30 Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου. Και συζήτηση αυτών 6 Οκτωβρίου. Ψηφοφορία και αυτή στις 6 Οκτωβρίου. Για να διότι καθήλυνα αρμόδια επιτροπή ψηφίσει στις 5 Νοεμβρίου. Θέλουμε να συντονίσουμε εργασίες μας με αυτή την επιτροπή. Σύντομο διάλειμμα μέχρι να έρθει ο κύριος Τρισέ. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τον έχει το λόγο του. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω ε, στην Επιτροπή για πρώτη φορά με αυτή, σε αυτή τη θητεία τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, η τελευταία συζήτησή μας ήταν 30 Μαρτίου και ε, η επόμενη για όσους ενδιαφέρονται ε, θα είναι ακόμη σε αρκετό καιρό οπότε όπως βλέπετε είχαμε μεγάλο κενό αλλά είχατε διάφορα σεμινάρια για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ανακαλύψατε πώς ε, λειτουργούμε. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω να παρουσιάσετε τα, ε, το θέμα σας και μετά θα προβούμε σε ερωτήσεις. Ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί ε, ε, μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Χρηματικών Υποθέσεων, χαίρομαι ιδιαίτερος που έχω την ευκαιρία σήμερα να ανταλλάξουμε απόψεις στην νέα σας θητεία. Είναι η 22η φορά που έρχομαι στην Επιτροπή αυτή. Είχαμε συχνές ακροάσεις που βοήθησαν να υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ε, του Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι θα βελτιωθούν οι σχέσεις αυτές σε μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική. Επίσης θα ήθελα τώρα να ε, επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Καταρχήν θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ε, αξιολόγησή μας της οικονομικής καταστάσεως στον ε, χώρο του ευρώ και θα ήθελα να αναφερθώ στα χρηματοπολιτικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της αποτελεσματικότητάς τους. Και επίσης για δεύτερη φορά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η αναμόρφωση της ε, δημοσιονομικής εποπτείας στην Ευρώπη ε, και στην κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Όπως βλέπετε έχουμε πλούσιο ρεπερτόριο και μετά θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Λοιπόν, η οικονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί από την προηγούμενη στο Κοινοβούλιο στις 30 Μαρτίου του 2009. Ο πληθωρισμός και οι σχετικές πιέσεις έχουν παραμείνει χαμηλές τους τελευταίους μήνες και ο πληθωρισμός έχει αναστραφεί αρνητικά το, κατά το καλοκαίρι λόγω της μειώσεως των τιμών πετρελαίου από πέρυσι. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός ήταν κάπως αρνητικός στο μείον 2% μετά από 0,7% ε, ε, τον Ιούλιο. Προβλέπουμε ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στο θετικό στους επόμενους μήνες και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Ελπίζουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμψει αλλά πολύ αργά. Ε, κίνδυνη κίνδυνη για πληθωρισμό είναι σαφής και ε, υπάρχουν δείκτες για αναμονή πληθωρισμού κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Ε, μετά από την ελεύθερη πτώση της οικονομικής δραστηριότητος ε, στο τέλος του περασμένου έτους, στο τομέα του ευρώ η οικονομία παρέμεινε σταθερή και μετά από τη σαφή μείωση που είχε αρχικά η οικονομική δραστηριότητα το δεύτερο δεύτερο τρίμηνο του 2009 μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο και προβλέπουμε ότι θα υπάρξει ανάκαμψη αλλά υπάρχει σαφής ε, ε, ε, αβεβαιότητα διότι από τη μια πλευρά υπάρχουν τα μακροοικονομικά προγράμματα κινήτρων και άλλα πολιτικά μέτρα για να βοηθήσουν την εμπιστοσύνη να ανακάμψει και η εξωτερική ζήτηση η οποία μπορεί να είναι ισχυρότερη από ό,τι προβλέπουμε. Υπάρχει όμως από την άλλη πλευρά η αρνητική ε, δράση μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και του ε, πιεσμένου ε, χρηματικού τομέα που μπορεί να αργήσει να ανακάμψει και υπάρχουν ακόμη ανισορροπίες. Επίσης η αξιολόγηση των χαμηλών πληθωριστικών πιέσεων μεσοπρόθεσμα καθορίζεται στην οικονομική μας ε, ανάλυση και ε, τονίζουμε ότι τα χρήματα και η ανάπτυξη ε, των πιστώσεων μειώνεται και προβλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ετήσια αύξηση των δανείων ε, μέχρι τον Αύγουστο. Ε, έχουμε όμως ε, μία πτώση παραγωγής και εμπορίου κατόπιν αυτού εφόσον η αύξηση των δανείων στις επιχειρήσεις έπεται της οικονομικής ανάπτυξης προβλέπουμε μία δυσχερή κατάσταση τους επόμενους μήνες συγχρόνως τα χαμηρά επιτόκια συνεχίζουν να οδηγούν σε χαμηλά επιτόκια δανεισμού το οποίο βελτίωσε τις καταστάσεις και τις συνθήκες χρηματοδοτήσεως και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει μία στήριξη στη ζήτηση για πιστώσεις στην ε, επόμενη περίοδο. Ε, γι' αυτό αξιολογεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα επιτόκια βάσει αυτών των στοιχείων και πρώτον έχουμε καλύψει τις ανάγκες ρευστών των τραπεζών με σταθερά επιτόκια δεύτερον έχουμε αναπτύξει τον κατάλογο των επιλεξίμων στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εγγύηση τρίτον έχουμε επεκτείνει τις περιόδους ε, ε, επαναχρηματοδότησης και τέταρτον ε, προσφέρουμε ρευστότητα σε διάφορα νομίσματα και ιδίως δολάριο για να καλύψουμε τις ανάγκες των τραπεζών του ευρώ να χρηματοδοτήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους που είναι σε δολάρια. Πέμπτον, έχουμε ξεκινήσει μία άμεση αγορά ομολόγων για να στηρίξουμε τις χρηματαγορές. Ε, Γενικώ τα μέτρα αυτά στηρίζουν ε, την ροή των πιστώσεων προς εταιρείε και τα νοικοκυριά ε, και μπορεί να επιτύχουν καλύτερα από ότι μόνο οι μειώσεις των επιτοκίων. Παρόλο αυτό όμως καταρχήν πιστεύω ότι δεν έχει λήξει η κρίση. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξουμε την ε, τα μέτρα μας. Κάποια στιγμή όμως θα χρειαστεί ε, να, ε, να βγούμε από την κρίση και θα πρέπει να υπάρξει στρατηγική εξόδου η οποία θα εφαρμοστεί διότι εάν θεωρούμε ότι τα άτυπα μέτρα ε, διακινδυνεύουν την οικονομική σταθερότητα, θα πρέπει να τα σταματήσουμε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, είναι πεπισμένη ότι πρέπει να ε, δρά όποτε είναι ανάγκη και ε, να υπάρχει θεσμική ανεξαρτησία για να μπορέσει να εφαρμόσει όποια δράση θεωρεί καλύτερα. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω αναφέρεται στη σχέση ρευστότητος και σταθερότητος τιμών, διότι ορισμένοι αναρωτιόνται αν το θαραλέο πρόγραμμά μας ε, μπορέσει να προκαλέσει πληθωρισμό στο μέλλον και πρέπει να σας εξηγήσω γιατί νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο φόβος Καταρχήν διότι η, η ρευστότητα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξηθεί αλλά δεν ε, οδήγησε σε μία αύξηση χρηματικών παραγόγων και ε, αυτό θα οδηγούσε υπομαλάς συνθήκας ε, σε ένα τέτοιο φαινόμενο για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως είπα και προηγουμένως η αύξηση των χρηματικών παραγόγων βασικό στοιχείο της διευρύνσεως της ρευστότητας στην αγορά είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και η τράπεζα ε, έχει όλα τα μέσα για να αποσύρει την στήριξη στη ρευστότητα εάν χρειαστεί. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι τα άτυπα μέτρα που λαμβάνουμε θα μειωθούν ε, σταθερά ε, όταν λήξουν εκτός και αν αποφασίσουμε να τα ανανεώσουμε. Ε, τώρα θα ήθελα να αφαιρθώ στο δεύτερο θέμα που είναι ο, ε, ε, η, η εποπτεία προληπτική εποπτεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η οικονομική κρίση έδειξε ότι το τωρινό σύστημα μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της συλλογικής συμπεριφοράς των παικτών της αγοράς και ιδίως ε, επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις των ε, χρηματαγορών και των στενών ε, δεσμών μεταξύ της προσφοράς πιστώσεως και της μακροοικονομίας συστημικοί κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να προκύψουν όταν τα χρηματοοικονομικά οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ελέγχουν τους κινδύνους τους κατά τρόπον ο, ο οποίος καλύπτει μόνο την προσωπική τους πρόπτικη. Ε, θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τα υπόλοιπα οικονομικά, τους υπόλοιπους οικονομικούς οργανισμούς και ε, η εποπτεία θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις αλληλοεπιδράσεις και τις ε, υποδομές των αγορών κατά τρόπον ώστε να συμβάλλει σε ένα κοινό καλό, δηλαδή στην ε, συστηματική οικονομική σταθερότητα. Σε συνδυασμό, η επίλυση των συστημικών κινδύνων θα πρέπει να ε, επιταθεί ιδίως εν ώψη της αυξανωμένης περιπλοκής των ε, παγκοσμίων ε, οικονομικών πράγμα το οποίο βοηθάει την, ε, από την τεχνολογική πρόοδο και γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσει να λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστηματικού Κινδύνου η σύσταση αυτού του Συμβουλίου είναι ε, ενδεδειγμένη και ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι συστάσεις που έχουν διατυπωθεί δεν πρέπει να παραμείνουν μόνο στα λόγια, θα πρέπει να υπάρξουν διατάξεις για να αναλάβουμε δράση ή να αιτιολογήσουμε γιατί δεν δράσαμε ε, για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε το Συμβούλιο αυτό, ιδίω θα πρέπει κανείς να εξηγήσει αν θέλει να συμμορφωθεί ή να εξηγήσει γιατί δεν το πράττει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό θα έχει πολύ στενέ σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα εκλέγουν τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Αυτού Συμβουλίου Εποπτείας όπως έχει προταθεί από την ομάδα Ντελαροζιέ και αναφέρθηκε από το Συμβούλιο και αποφασίστηκε στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ε, και υιοθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Όπως σας είπα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι έτοιμη να θέσει όλους τους ε, αναγκαίους πόρους στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, του Εποπτικού αυτού Συμβουλίου σε συνεργασία με τις 27 κεντρικές τράπεζες. Ε, η νέα κατάρτιση του Εποπτικού Συμβουλίου και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκεί θα πρέπει να έχει σταθερές βάσεις και θεσμικές και νομικές ε, για να μπορέσει η τράπεζα να συμβάλλει θετικά εις ε, την κατάρτιση του Εποπτικού Συμβουλίου και ε, να ε, επιτρέψει την μακροοικονομική εποπτεία με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Δεν μπορεί δηλαδή η Ευρώπη να παραμείνει αδύναμη και να μην μπορέσει να καλύψει και να ανταποκριθεί στους κινδύνους οι οποίοι παρουσιάσονται. Επί του θέματος αυτού θα απαντήσω σε ερωτήσεις όταν θα μου τις θέσετε και θα ήθελα να σας πω κυρία Πρόεδρε ότι από ό,τι βλέπω πολλές από τις πρωτοβουλίες έχουν, έχουν προκληθεί εδώ από τις συζητήσεις αυτής της Επιτροπής. Τέλος όσον αφορά την, ε, τον απολογισμό. Ε, το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Εποπτικού Συμβουλίου θα είναι πολύ στενή δεν σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να συγχωνευτούν οι εργασίες αναφοράς προς την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο. Ο στόχος μας είναι να παραμείνουν δύο διαφορετικές ενέργειες ε, διότι υπάρχει σαφής εντολή και όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα το, η συνθήκη στο άρθρο 105.1 λέει ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι να διατηρήσουμε σταθερότητα τιμών και όσον αφορά την δημοσιονομική σταθερότητα η συνθήκη μιλά για μία σύμβολη στο άρθρο 105.5 λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να συμβάλλει στη σταθερότητα του δημοσιονομικού συστήματος και αυτό το έργο περιλαμβάνει ότι ε, το, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να ε, παρουσιάσει τις προτεραιότητες ε, και τον εντοπισμό αυτών των κινδύνων και να προειδοποιεί όταν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ο οποίος φαίνεται σημαντικός. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για το ότι καταστήσατε σαφές ότι δεν προτίθεστε να συγχωνεύσετε αυτές τις δύο εκθέσεις. Είμαστε ευγνώμονες για αυτή την επιβεβαίωση από πλευρά σας. Και περνάμε τώρα στις ερωτήσεις. Υπό τους ίδιους κανόνες όπως θεσπίστηκαν και στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία μας, κάθε ερωτών θα έχει 1,5 λεπτό στη διάθεσή του. Μετά εσείς κύριε Τρισέ θα έχετε 3,5 λεπτά να απαντήσετε. Αυτό θα τηρήσουμε και αν το τηρήσουμε θα μπορέσουμε τις περισσότερες ερωτήσεις να τις καλύψουμε. Ξεκινάμε με την ομάδα του ΕΛΚ. Ο Ζαν Πολ Γκοζές παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Για μία ακόμη φορά με χαρά σας υποδεχόμαστε εδώ. Μας διαφωτίσατε σε σημαντικά θέματα και από την πλευρά μου είμαι ευτυχή που ξαναβλέπω, διότι αυτό σημαίνει ότι συνεχίζω τη θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελευταία φορά που συζητήσαμε, σα είχα θέσει ένα ερώτημα που αφορούσε τον πληθωρισμό. Επιτρέψτε μου να επανέλθω, είναι μανία δική μου κι αυτή. Κάποιες χώρες έχουν ένα χρέος πάρα πολύ μεγάλο όσον αφορά την Ευρώπη. Έχετε την νομισματική ζώνη, την ελεγχόμενη, δώσατε κάποια στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη, αλλά όλος ο κόσμος ε, δεν αντιλαμβάνεται ε, την εξουσία που έχει η Κεντρική Τράπεζα, δεν βασίζεται στην Κεντρική Τράπεζα και σε άλλες χώρες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχουν υπερβολικά χρέη και αυτά τα χρέη ίσως μπορεί εν μέρη μέσω νομισματοποίησης ε, μπορούν να απορροφηθούν ή να αφήσουν ανεξέλεκτες συστημές. Αν γίνει κάτι τέτοιο, ποια θα είναι η απάντηση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λαμβάνεται υπόψη της διατάξης των συνθήκων, τον ενεργό ρόλο της τράπεζας όσον αφορά τη διατήρηση των τιμών, άλλο σχόλιο όσον αφορά το Συμβούλιο του Συστημικού Κινδύνου, το Κοινοβούλιο επελήφθη του θέματος και θα σας πω ότι θα φροντίσουμε ούτω ώστε οι δικές σας ανησυχίες επίσης να είναι και δικές μας και να μεταφραστούν ε, σε κείμενα τα οποία θα μας υποβληθούν τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερος που σας ξαναβλέπω, μαζί και μερικούς συναδέλφους σας. Είναι σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι παρατηρώ και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση απόψεων Πιστεύετε ότι χωρίς σταθερότητα τιμών μέσω μακροπρόθεσμα ε, θα έχουμε πολύ αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα. Είχατε υποθέσει ότι υπάρχει πληθωρισμός από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού όταν θέσατε το ερώτημα. Δεν είναι πρόθεση της Federal Reserve, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, να κάνω αυτά που είπατε και είναι πεπισμένη η Federal Reserve που και εμείς, ανεξάρτητα από την εντολή που έχουμε, να έχουμε σταθερότητα, να επιβάλλουμε τη σταθερότητα τιμών, κάτι που απαιτούν οι συνθήκες και σας λέω εν είδη απαντήσεως ότι θα εφαρμόσουμε τις συνθήκες. Όλες οι συνθήκες, τίποτα παρά τη συνθήκη. πρώτο ρόλο έχουν η έχει η σταθερότητα των τιμών και βασιστείτε πάνω μα. Είμαστε σημείο αναφοράς εμπιστοσύνη και σταθερότητα. εμπιστοσύνη λέω, διότι οι συμπολίτε μας πολύ συχνά μας λένε ότι ανησυχούμε μέσω μακροπρόθεσμα και πιστεύω ότι μπορούμε να τους καθησυχάσουμε. Είμαστε ακριβώς εκεί για αυτό το σκοπό, για να εξασφαλίζουμε σταθερότητα τιμών. Εάν δεν εξασφαλίζαμε σταθερότητα τιμών και αν αυτό ίσχυε και τι δύο πλευρές του Ατλαντικού, είναι μια υπόθεση που αποκλείω εντελώ, αλλά φανταζόμαστε τώρα. Λέμε, φανταζόμαστε, τι θα γινόταν. όλε οι αγορέ στο επιτόκιο των αγορών μέσο και μακροπρόθεσμα 2, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 30 χρόνια, 50 χρόνια διότι κάποιες κυβερνήσεις δανείζονται για 50 χρόνια το μελλοντικό πληθωρισμό και θα ενσωμάτωναν το μελλοντικό πληθωρισμό στα επιτόκια τους της αγοράς. Οπότε το χρέος αντί να μειώνεται σταδιακά λόγω πληθωρισμού θα αυξανόταν, θα αυξανόταν, θα αυξανόταν και η φούσκα, ο πομφόλιγας αυτός θα μεγεθυνόταν συναρτήσει των επιτοκίων της αγοράς που θα συμπεριελάμβανα τον πληθωρισμό. Εγγυόμενοι τώρα τη σταθερότητα των δημών, εμείς της Κεντρικής Τράπεζας βοηθούμε να ξεφύγουμε από μια τέτοια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αδιαμφισβήτητα από πλευράς δημοσιονομικών είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σημείωσα δεόντως το σχόλιο σας για το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορούμε να έχουμε άκρος καρποφόρο διάλογο. Παρατείνεται αυτός ο διάλογος άλλωστε στον οποίο συμμετείχατε πριν από αρκετούς μήνες, διότι θυμάμαι πάρα πολύ συχνά από το Κοινοβούλιο απευθυνόταν το αίτημα αυτό από την Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να συναντώμαστε πιο συχνά και να συμμετέχουμε, ε, ε, να υπάρχει πιο συστημικός, συστηματική συμμετοχή μάλλον στο Συμβούλιο αυτό του συστημικού κινδύνου. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ο Γκέι Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξαιρετικά αντιμετώπισε το θέμα του πληθωρισμού όχι όμως σε σχέση με το asset inflation. Σας είχα ρωτήσει ε, επίμονα και πριν από δύο χρόνια για αυτό το θέμα του asset inflation για τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα για την Ιρλανδία και τις επιπτώσεις αυτού του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται ότι δεν είχε την δύναμη να δράσει, ήταν αδύναμη. Και αυτό μπορεί να συμβεί και με άλλες χώρες έπρεπε να είχε γίνει κάτι ή τουλάχιστον σε σχέση με το asset inflation στον ε, εναρμονισμένο δείκτη για τις ε, ε, δαπάνες καταναλωτή μπορούσε να έχει ανιχνευθεί και να έχει γίνει κάτι σε σχέση με την Ιρλανδία, σε σχέση και με τις επιπτώσεις που είχε αυτό εκεί. Έχετε κάποιες ανησυχίες ίσως για την προσέγγιση που υιοθετείτε για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος από πλευράς Ιρλανδίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είσαστε πραγματικά θα έλεγα συνεπέστατος ε, παρακολουθώντας αυτό το θέμα και για εύλογους λόγους. Επιτρέψτε μου να πω ότι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξετάζουμε και βλέπουμε το τι ευθυγραμμίζεται με την κυρίως εντολή μας ε, για την διασφάλιση της ευημερίας ε, για το σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στο ευρώ. Είναι λοιπόν για κάθε χώρα δική της υπόθεση το να λάβει υπόψη ότι εμείς βελτιστοποιούμε την νομισματική πολιτική στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Και αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι όποιες ανομαλίες υπάρχουν διορθώνονται από τα εθνικά μέσα και με την φορολογική πολιτική και την νομισματική πολιτική που ακολουθείται και το είδος της προληπτικής αντιμετώπισης συνετής διαχείρισης prudential όπως και από τον πυλώνα της Βασιλείας 2 ρυθμιστικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο για επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Ανέφερα κάποια εργαλεία, κάποια μέσα που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο φυσικά συμμετέχουν ε, οι ε, κεντρικοί τραπεζίτες ε, των κρατών μελών και που ενεργά και με κάθε στένος συμμετέχουν, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω το ότι αν λοιπόν η ιδέα είναι ότι δεν λάβαμε παρκώς υπόψη ή δεν ασχοληθήκαμε επαρκώς με την λήψη αποφάσεων για την, στοχοθετημένα για την πρόληψη τέτοιων πομφολίγων και να υπενθυμίσω ότι ασκήθηκαν έντονες επικρίσεις το 2004 κατά την αρχή του 2004 διότι δεν μειώναμε τα επίπεδα των επιτοκίων όταν ζητήθηκε και ερωτήθηκε σε σχέση με το 2% να πάμε στο 1% είπαμε όχι εμείς αντιμετωπίσαμε με σθένος το θέμα αυτό ασκήθηκαν έντονες επικρίσεις σε σχέση με τα επίπεδα αυτά. Στην συνέχεια βρισκόμαστε στο 2% και θεωρήθηκε ότι έπρεπε να υπάρξει και μία αύξηση. Και στις δύο περιπτώσεις ασκήθηκαν επικρίσεις από εκείνους που έβλεπαν μόνο τα θέματα οικονομικών αναλύσεων. Αλλά επίσης εμείς εξετάζουμε και τα θέματα νομισματικών αναλύσεων και την εξέλιξη των νομισματικών συνιστοσών με πιστώσεις και μέσω πιστώσεων και για την ε, διαμόρφωση των assets prices. Θα έλεγα λοιπόν ότι μεταξύ της συγκυρίας και των θεμάτων των κεντρικών τραπεζών είμαστε εμείς αυτή η κεντρική τράπεζα λόγω του διπυλωνικού συστήματος που υιοθετούμε οικονομικής ανάλυσης και νομισματικής ανάλυσης είμαστε εμείς η κεντρική τράπεζα που προσπαθεί να ενσωματώσει στο μέγιστο το δικό σας μέλημα και την ανησυχία σας που είναι σημαντικότατο θέμα φυσικά επιτρέψτε μου να πω ότι το θέμα αυτό από πλευράς ακαδημαϊκού υιοθετείται ε, η βέλτιστη προσέγγιση γίνεται μεγάλη προσπάθεια να το, να το αντιμετωπίσουμε. Προσεγγίζουμε θα έλεγα ίσως με αυτόν τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο να επανενσωματώσουμε αυτό το μακροπρόθεσμο μέλημα το οποίο έχετε στις ε, ενέργειές μας. Και θα έλεγα ότι εδώ όσον αφορά την μακροπρόθεσμη, με μεγάλο μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα της νομισματικής σταθερότητας, δεν υπάρχει κάποια αντίφαση σε σχέση με τον δυναμισμό των νομισματικών παραγόγων. Νομίζω ότι μπορεί αυτό να θεωρηθεί αλληλοσυμπληρούμενο. Ευχαριστώ. Χωσέ Μανουέλ, είσαι έτοιμος? για την ερώτησή σου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρεις παρατηρήσεις ε, εντάχει με την εξή ε, στην συνέχεια ερώτηση. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και που μεγάλη, με μεγάλη χαρά τον ξαναβλέπω σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία πάλι επισήμανε ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη όμως η αλήθεια είναι ότι οι πιστώσεις δεν φτάνουν στην πραγματική οικονομία και δεν έχουμε την πραγματική επίπτωση που αναμέναμε. Στην αρχική παρέμβαση θεώρησε υπεύθυνο για αυτή την έλλειψη, απουσία πιστώσεων, την έλλειψη ζήτησης μου φαίνεται ότι δεν είναι αυτή η ας το προσέγγιση πολλών επιχειρήσεων και πολλών οικογενειών στη χώρα μου που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις επειδή οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια και πιστώσεις. Και σε σχέση με αυτό θα ήθελα να ξέρω το, το Ευρωβαρόμετρο, οι δικές σας φυγμομετρήσεις ε, επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη των ε, ε δανειοληπτών ε, των πολιτών μας. Δεύτερον, σε σχέση με την σωστή θεωρία θα πρέπει να ξεκινήσουμε να ενεργούμε με τον τρόπο εκείνο που θα αποκαταστήσει τα πράγματα σε σχέση με τον ασθενή. Και ο διοικητή τη Κεντρικής Τράπεζα θεωρεί ότι πολλά από τα μέτρα μη στάνταρτ ή ανορθόδοξα θα μπορέσουν να απαλληθούν αφεαυτών, δηλαδή αφεαυτών θα απαλληφθούν και καθώς επίσης και η αύξηση των ε, ε, συμπληρωματικών μέτρων που θα δέχεται η Κεντρική Τράπεζα. Δεύτερον, οι προθεσμίες για τις οποίες συζητήσαμε ε, εκτενώς για την αποκατάσταση πιστώσεων. Έξι μήνες είναι πολύ πιεστική προθεσμία ε, επίσης για άλλες ε, προθεσμίες επανεξετάζει αυτά τα θέματα η Κεντρική Τράπεζα ή αυτά τα δύο θα έχουν σταθερό μόνιμο χαρακτήρα. Η τρίτη και τελευταία τώρα παρέμβαση ως ερώτηση για το συστημικό κίνδυνο. Η Κεντρική Τράπεζα θα ε, υποβάλει συστάσεις Πώς θα διασφαλίσετε ότι οι χώρες θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να υιοθετήσουν αυτές τις συστάσεις. Θα υπάρξει κάποια μορφή ε, κυρώσεων ε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ε, θα υπάρξει μια ήπια, ας το πω έτσι, προσαρμογή. Τι θα γίνει από πλευράς αυτής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εύχομαι και συγχαρητήρια σε σχέση με τις προσπάθειες. Thank you Ευχαριστώ. Οι ερωτήσεις σας είναι πολύ σημαντικές. Όσον αφορά την κατανομή των πιστώσεων, είναι προφανές ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο διαπιστώνουμε τους πρόσφατους αριθμούς ότι οι πιστώσεις ε, ε, δεν ε, αναπτύσσονται είναι διότι η πραγματική οικονομία όπως είπατε και εσείς έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ και συρρυκνώθηκε και η ζήτηση. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, τις οποίες εξετάσαμε ιδιαιτέρως, είδαμε ότι το 77% της αιτήσεως πιστώσεων οδήγησαν σε θετική αντίδραση 12% όχι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα της κατανομής λειτουργεί σωστά και δεν μπορώ να σας πω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, αλλά προφανώς ο ρόλος των τραπεζών σε μια οικονομία αγοράς πρέπει ορισμένες φορές να είναι να αρνούνται ε, και αυτό μας φαίνεται φυσιολογικό αλλά πρέπει 77% που είναι ε, θετικό θα οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα ε, εν ευθέτω χρόνο αλλά η ζήτηση ε, ευθύνεται για την έλλειψη δυναμισμού την οποία διαπιστώνουμε ως προς, ως προς τις πιστώσεις. Όσον αφορά τα άλλα μέτρα τα οποία ανέφερα, όπως σας είπα υπάρχουν πέντε ατυπικά μέτρα. Καταρχήν, ε, οι κεντρικές τράπεζες θα ξεκινήσουν μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση έξι μηνών μέχρι ενός έτους. Ήμασταν και οι πρώτοι οι οποίοι έχουν ε, διευρύνει την επιλεξιμότητα των εγγύσεων και οι πρώτοι οι οποίοι έχουν διαγνώσει ε, την κατάσταση δηλαδή ήδη από τον Αύγουστο του 2007 είχαμε δηλώσει ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και τελικά δικαιωθήκαμε ατυχώς. Βεβαίως δεν πρέπει να διακινδυνεύσει η σταθερότητα των τιμών ε, το οποίο είναι βασικό στοιχείο για τους Ευρωπαίους ε, για να μπορέσει να υπάρχει συστηματική ανάκαμψη. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι μελλοντικές ε, οι μελλοντικές προσδοκίες ε, πληθωρισμού ενσωματώνονται στις, ε, στα τωρινά μέτρα οπότε πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε μέτρα για να μπορέσουμε να αποδώσουμε, να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τηρημών και δεν πρέπει μόνο να κοιτάξουμε τι κάνουμε τώρα αλλά και τι θα πράξουμε εν ευθέτω χρόνο. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο στόχος της ESRB θα είναι να εντοπίσει τον κίνδυνο ε, και να διατυπώσει συστάσεις δεν θα υποκαταστήσει τις διάφορες αρχές για να λάβει αποφάσεις διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως σας είπα. Λοιπόν. Ο κύριος ε, Σάντσες Πεσέδο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα ο ίδιος να ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία εδώ ανάμεσά μας του κυρίου Τρισέ και να εκφράσω επίσης την εξής άποψη η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι πολύ καρποφόρο, πολύ γόνιμο για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και εγώ θα αναφερθώ σε δύο ερωτήσει. Η πρώτη αναφέρεται πιο εξειδικευμένα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δεύτερη στην μακροοικονομική επιτήρηση. Φαίνεται ότι στην οικονομική κρίση το πιο οξύ, το πιο έντονο τμήμα πέρασε και χρειάζεται τώρα η ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης και η ε, κατάσταση των ανισορροπιών. Και εδώ και περίπου ένα μήνα ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μπερνάκε της ε, ε, Κεντρικής Τράπεζας τον είπε, είπε δεν θα γίνει κάτι τέτοιο μέχρι ότου μπορέσει να ανοίξει ε, τις πύλες του η πίστοση, τις πύλες της η και εδώ αφορά αυτό άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ε, δανειοδότηση των τραπεζών. Πλήττονται άμεσα λοιπόν σε σχέση με την ε, χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Υπάρχουν αυξημένες ε, ανάγκες και φαίνεται εδώ ότι σε σχέση με την τραπεζική πιστο, τη διάθεση πιστώσεων από τις τράπεζες πρέπει να αποκατασταθούν τα πράγματα. Πότε μπορεί να γίνει αυτό. Δεύτερη ερώτηση με την μακροεπιτήρηση. Πιθανότατα με την χρηματοοικονομική κρίση υπάρχει ανάγκη και το έχουμε αναγνωρίσει μια επιτήρηση ε, πέρα από τα θεσμικά όργανα με ένα συστημικό χαρακτήρα. Είναι προφανέ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τι συνθήκε έχει λόγο να εκφράσει και θα πρέπει να διαβουλεύεται επ' αυτού του θέματο και να γνωμοδοτεί. Ενδιαφερόμαστε άμεσα να γνωρίζουμε αν αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των ε, συστημικών κινδύνων, για τις ε, εξουσίες που έχει επαρκούν ε, για να αντιμετωπιστεί η εντολή σε σχέση με την χρηματοοικονομική κρίση, σε σχέση με προειδοποιήσεις για παράδειγμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι συστάσεις αυτές είναι επαρκείς, δεν πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του οργάνου σας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συστημικοί κίνδυνοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα προτείνατε μια ειδική δομή μέσα από αυτό το Συμβούλιο και πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί η διεθνή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, πράγματι, στη δική μας ανάλυση, από το τέλος του δευτέρου τριμήνου αυτού του έτους, είμαστε στο τέλος της ελεύθερης πτώσης της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Πτώση που ζούμε από τα μέσα Σεπτεμβρίου πέρσι. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα γεγονός που δημιούργησε δραματικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Βγήκαμε από την περίοδο ελεύθερης πτώσης. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να παραμείνουμε προσεκτικοί. Όπως ξέρετε, έπρεπε να ανεριθούν προς τα πάνω οι προβλέψεις και όσον αφορά το μέσο όρο για φέτος και του χρόνου, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι πολύ αρνητικό το τρέχον έτος, ακόμα και αν είναι 0,5% καλύτερα τα πράγματα από ό,τι προβλεπόταν αρχικά και το ίδιο και για τον επόμενο χρόνο. Ελαφρά θετική εξέλιξη, πολύ κοντά στο 0. Ο δρόμος χωματόδρομος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, επιφυλακτική, να επαγρυπνούμε, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε είναι. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι σημαντικότατο στομέα αυτές οι επιχειρήσεις δημιουργούν τις θέσεις απασχόρες που χρειάζονται και παρακολουθούμε προσεκτικότατα τα όσα συμβαίνουν σε αυτό το τομέα. Έχουμε επικεντρωθεί, όπως ξέρετε, όλο, όλα τα μη συμβατικά μέτρα μας στις τράπεζες, διότι θεωρήσαμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε πιστώσει μόνο μέσω των τραπεζών, όχι μέσω των αγορών. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό να επικεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα ε, στο δίευλο αυτό των τραπεζών. Διαφορετική προσέγγιση με τις ΗΠΑ αλλά εξηγείται από την κατάσταση την ευρωπαϊκή και από την μέρημνά μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εξηγούμε στις τράπεζες, κοιτάξτε τι κάνουμε για σας. Ό,τι κάνουμε είναι για σας μη συμβατικά μέτρα και το επίπεδο των επιτοκίων που επιβάλλουμε. Όλα αυτά γίνονται όχι για σας αλλά για την πραγματική οικονομία, για να συμμετέχετε εσείς ένεργα στην ανάκαμψη. Που είναι κοινός μας στόχος και πρέπει να πω ότι σε αρκετές περιπτώσεις λέμε στις τράπεζες. Κοιτάξτε, αν θέλετε κι άλλο κεφάλαιο, εποφεληθείτε από τα χρήματα που έθεσε στο αποθεματικό η κυβέρνηση σαν νέο κεφάλαιο. Τη στιγμή που μιλώ εκτιμούμε ότι 55% του κεφαλαίου που είχε προσημειωθεί από τις κυβερνήσεις για ενδεχόμενη ανακεφαλοποίηση έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά 45% δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Οπότε υπάρχουν δυνατότητες και πάντα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης προσφυγής στην αγορά. Τούτων λεχθέντων. Το μήνυμα προς τις τράπεζες είναι σαφές. Κάντε τη δουλειά σας. Τώρα, όσον αφορά το συστημικό κίνδυνο και το σχετικό συμβούλιο, συμφωνώ με το σχόλιο σας. Πράγματι, είναι εξαιρετικά σημαντικό η συνέχεια να είναι άριστα διοργανωμένη και ποια έννοια ακολουθούμε. Ισχυρή πυθό, ηθική πυθό όσον αφορά το Συμβούλιο Συστημικού ε, Κινδύνου, δεν χρησιμοποιούμε άλλες δυνατότητες. Παίρνουμε τα πράγματα ως έχουν. Το έλεγα, οι συνάδελφοί μου και εγώ είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά σε αυτό το Συμβούλιο. Δεν είναι το ECD. Τόσο φορές κάνει αυτά που είπε στην αγωγή. Συμβάλλει στην επιτυχία του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και υπάρχει πολύ στενή διασύνδεση με τι εργασίε του Συμβουλίου Κινδύνου. Δεν πρέπει να συγχαίουμε όμω τι ευθύνε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τι ευθύνε του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Μα ξεφεύγει κάπω ο χρόνο, καθυστερούμε. Ο Ρόμπερτ Μπέγκελ έχει το λόγο. Γκέμπελ, συγγνώμη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πολύ που σα ξαναβλέπω και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπαιξε πολύ σωστά το ρόλο της γιατί επέτρεψε να αναχρηματοδοτηθούν οι τράπεζες ε, και παρόλα αυτά όμως ε, οι δράσεις αυτές και η προσφορά πιστώσεως δεν βοήθησαν τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις το είπατε και μόνοι σας. Μία αύξηση τον ε, Αύγουστο κατά 0,1% και όπως το είπε και ένα συνάδελφος δεν μπορεί χωρίς αύξηση των πιστώσεων να υπάρχει ανάκαμψη. Όλα τα μέσα τέθηκαν στις τράπεζες σε τι βοήθησαν. Νομίζω ότι οι τράπεζες με τα λεφτά αυτά αγόρασαν, ε, ε, ε, αγόρασαν χρεόγραφα. Δεν μπορείτε εσείς να χρηματοδοτήσετε τις κυβερνήσεις τα δώσατε εύκολα λεφτά στις τράπεζες και νομίζω ότι αυτές οι πιστώσεις και η χρηματοδότηση ε, πέτρεψαν σε τράπεζες να κερδοσκοπήσουν στις ε, ε, νομισματαγορές. Μήπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να εφαρμόσει πιο περιοριστικά κριτήρια για τις χρηματοδοτήσεις ιδίως ε, που θα έχουν ε, πολύ μακριά προθεσμία λήξεως. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Θα σας έλεγα ότι το μήνυμά μας προς τις τράπεζες πάντοτε ήταν αυτό το οποίο προανέφερα. Δηλαδή ότι εμείς αυτά που κάνουμε δεν τα κάνουμε τόσο για την νομισματική πολιτική όσο και για τα άτυπα μέτρα για τα ωραία σας μάτια αλλά για να κάνετε το, τη δουλειά σας σωστά δηλαδή να χρηματοδοτήσετε την οικονομία όταν ένα μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν θετικά τα μέτρα αυτά δεν μπορώ να σας πω ότι η διαπίστωση είναι τόσο κακή όσο εσείς διατείνεστε. Αυτό όμως που κατάλαβα από την ερώτησή σας είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς στο μήνυμά μας. Είναι το μήνυμα των κεντρικών τραπεζών, διότι όντως κάνουμε πολλά και ε, ε, όπως, ε, όπως συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συμβαίνει και στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και διεθνώς και στις κυβερνήσεις ακόμη οι οποίες αποφάσισαν και έπρεπε να αποφασίσουν εμείς τους ζητήσαμε και τους είπαμε ότι έχουμε πρόβλημα συστηματικής ρευστότητα σημαντικό πρέπει να το επιλύσουμε δεν μπορεί να υπάρχει συστηματική φερεγγιότητα διαφορετικά γι' αυτό και η κεφαλαιοποίηση η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δανειό δότησης και ε, η βοήθεια για τα τοξικά ε, χρεόγραφα ε, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει όμως μια οικονομία ανοιχτής αγοράς και εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τις τράπεζες. Είμαστε σε μια οικονομία αγοράς όπου πρέπει να υπάρχουν αποκεντρωμένες αποφάσεις, διαφορετικά δεν πάμε καλά. Αλλά η ε, ηθική πυθός θα πρέπει επίσης να επηρεάσει και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ, ο κύριος Φιν. Κύριε Πρόεδρε, Συμφωνώ με την άποψή σας ότι όντως υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται και σαν ελεύθερος δημοκράτης από τη Γερμανία πρέπει να σας πω ότι είμαι αισιόδοξη ε, ιδίω λόγω των αποτελεσμάτων των εκλογών στη χώρα μου και γι' αυτό ε, προσβλέπω θετικά και αισιόδοξα προς το μέλλον ο κύριος ο Λόρδος Τέρνερ της ε, FSA έκανε διάφορες ε, ε, ιδιόρυθμες προτάσεις για το πώς μπορεί κανείς να ενισχύσει το χρηματοοικονομικό σύστημα και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες διάφορα ποσοστά τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν. Πιστεύετε εσείς για την εποπτεία ότι θα πρέπει ε, η Επιτροπή αυτή να εξετάσει τις προτάσεις που διατυπώνονται ή αυτό είναι καθήκον ενός εποπτικού οργάνου και εσείς απλούστατα ε, διαπιστώνετε την ανάγκη εποπτείας. Επίσης ήθελα να σας πω δεν θα ήταν καλό να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα καταγραφής των πιστώσεων και των κινδύνων ώστε να μπορεί κανείς πολύ γρήγορα να δει από πού και πώς ε, υπάρχουν κίνδυνοι ε, πράγμα το οποίο τώρα επιτυγχάνεται μόνο με πολύ δύσκολο και πόδινο τρόπο όπως ξέρετε ε, καλύτερα από οποιονδήποτε το θεσμικό όργανο που αντιπροσωπεύω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαντά σε όλες τις ευαισθησίες ε, σε, ε, στα εκατομμύρια των συμπολιτών μας σε εκατοντάδες εκατομμυρίων των συμπολιτών μας είναι λοιπόν βασικό να να πιστεύουμε ότι το μελλοντικό εποπτικό συμβούλιο ε, θα πρέπει να καταρτιστεί ε, με διαδικασίες συνένεσης γιατί πολλές ιδέες για την εποπτεία στην ε, ασφα... στις ασφάλειες στις αγορές και τα λοιπά είναι απαραίτητες και γι' αυτό και θεωρώ ότι η εποπτική αρχή της Επιτροπής της Βασιλείας ε, και το Pittsburgh σε επίπεδο αρχηγών κρατών ε, μπορούν να συμβάλλουν στην ε, ε, αύξηση της εποπτείας των τραπεζών διεθνώς με κάθε τρόπο και σε όλες τις χώρες ακόμη και στις αναδιόμενες χώρες διότι είδατε ότι το Pittsburgh στήριξε την κίνηση αυτή προς καλύτερη εποπτεία. Πιστεύω λοιπόν ότι το εποπτικό αυτό συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μακροπρόθεσμα μέτρα προβλέψεων για να μπορέσει να βελτιώσει τις ε, ενέργειές τους και να αναλάβει την ευθύνη ε, των ε, αρχών για την μικροαξιολόγηση του κινδύνου διότι όπως ξέρετε υπάρχουν οι κεφαλές των ε, τριών ε, θεσμικών οργάνων στην Ευρώπη. Δεν είναι όμως εύκολο αυτή τη στιγμή να προεξοφλήσουμε τη μέλη γεννήστε. Δεν μπορούμε ε, παρά μόνο να κάνουμε αυτό που μας ζητούν και αν είναι αναγκαίο να προβούμε σε μία έγκαιρη προειδοποίηση και να διατυπώσουμε προτάσεις όπως αυτές τις οποίες ε, ε, ανέφερε ο κύριος Τέρνερ. Βέβαια, ε, εγώ δεν τάσομαι υπέρ κατά, απλούστατα πιστεύω ότι υπάρχει γενική συνένεση ότι ναι μεν υπάρχουν οι απαιτήσει της Βασιλείας 2 ή ε, για τις ανάγκες κεφαλαίου ή τους κινδύνους που έχουν καθοριστεί πέραν αυτού όμως πρέπει να ε, εξετάσουμε το ε, ποσοστό μόχλευσης διότι διαφορετικά θα πρέπει να υπολογίσουμε πού βασιλεύει ο κίνδυνος και ορισμένες φορές το ποσοστό μοχλεύσεως μπορεί να στρεβλωθεί. Ε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι θα συνεχίσουμε να ε, εργαζόμαστε στεναρά επί του θέματος αυτού. Κύριο Σέπεν. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υπό μαλά συνθήκας προσπαθούμε να διευκρινίσουμε τις της προηγούμενης κρίσης και ε, για να μπορέσουμε ε, να αξιολογούμε τα συστήματα σωστά. Θα ήθελα να ξέρω το Συμβούλιο αυτό το εποπτικό πόσα, πόσο μεγάλο θα είναι, πόσα μέλη θα έχει, πώς θα αποφασίζεται αν υπάρχει συστηματικός κίνδυνος διότι ε, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα ξέρω ότι ε, θεωρούν ότι οι αμερικανικές ε, ε, υποθηκευτικές τράπεζες δημιούργησαν το πρόβλημα. Πώς θα το αποφύγουμε λοιπόν και τι εξουσία θα έχει αυτό το Συμβούλιο, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές τους. Υπάρχουν χώρες που είναι στο ευρώ και χώρες που δεν είναι. Για να πάρω παράδειγμα κατά τύχη το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να πει η εποπτική αρχή αυτή στην Αγγλία δεν λειτουργείτε σωστά πρέπει να κάνετε αυτά που εμείς σας υπαγορεύουμε ε, διότι εδώ υπάρχει ένα κείμενο το οποίο λέγει και θα το διαβάσω αγγλικά ε, έχουμε δικαίωμα να λάβουμε ε, σαν τελευταία καταφυγή ε, κανόνες οι οποίοι θα εμποδίσουν τις τρέβλες της αγοράς. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μου πείτε σε απλά αγγλικά τι σημαίνει αυτό το οποίο μας διαβάσατε. Καταρχήν, μου ζητάτε χωρίς ε, να είστε μεταξύ αυτών ε, που μας κατακρίνουν να σας πω ότι είμαστε στη διάθεση της Ευρώπης για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτού του συστηματικού κινδύνου. Μη μου θέτετε λοιπόν ερωτήσεις που θα έπρεπε να θέσετε στην Επιτροπή ενδεχομένως στο Συμβούλιο ή όπου υπάρχει συναπόφαση. Για να είμαι σαφής. Αυτό που αντιλαμβάνουμε είναι το εξής Καταρχήν έχετε τους ε, ε, διοικητές των 27 κεντρικών τραπεζών και γι' αυτό υπάρχει ένα σύστημα ESCB δηλαδή οι 27 αρχές Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας. Έχουμε λοιπόν τους διοικητές, τον διοικητή και υποδιοικητή διοικητή της ε, Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας ε, και τους μακρο επιτηρητές όπως είναι η Επιτροπή. Αυτοί θα συζητήσουν σαν μια Επιτροπή Σοφών τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, ε, χρηματοοικονομικής πολιτικής και βάσει της σοφίας τους ε, για να υπάρξει μία μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη θα διατυπώσουν προτάσεις. Δεν θα αντικαταστήσουν τις εμπλεκόμενες αρχές είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Δεν πρόκειται να τις υποκαταστήσουν αλλά θα αναφερθούν σε εσά και θα αποφασίσουν εάν ή όχι θα δημοσιοποιήσουν τις συστάσεις αυτές και στη συνέχεια αυτές οι σοφές συστάσεις θα μπορέσουν να ε, συνοδευτούν με δράσεις. Αλλά όπως σας είπα και πάλι δεν θα αντικαταστήσουμε αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν τις αποφάσεις. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραίο να σας ξαναβλέπει κανείς κύριε Τρισέ. Είναι ωραίο το ότι είσαστε πάλι ανάμεσά μας. Μία ερώτηση θα είχα, η οποία αναφέρεται στα εξαιρετικά μέτρα, έκτακτα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εσείς σε σχέση με ε, ασφάλειες ε, που δεχθήκατε, που πολλές φορές θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει, θα με ενδιέφερε είδα την ετήσια έκθεση 2008 από πλευρά σας. Πόσο μεγάλο είναι το τμήμα των μη καλυμμένων asset securities σε σχέση με το 2009, σε σχέση με όλα τα assets που από ιδιωτικές τράπεζες εγκρίνατε ή δεχθήκατε. Και σας ρωτώ επίσης ποιες επιπτώσεις απορρέων πιστεύετε εσείς για τις τράπεζες, αν αυτοί οι κίνδυνοι και αυτές οι ασφάλειες ε, πρέπει να ε, αποσυρθούν τα έκτακτα μέτρα δηλαδή όταν θα λήξουν και δεν θα ισχύουν πλέον και δεν θα καλύπτονται αυτές οι ασφάλειες. Θα με ενδιαφέρει για τη σταθερότητα και τη φερεγγιότητα των τραπεζών όταν αυτό το μέτρο ακυρωθεί. Και εν τέλει, δεδομένων των μεγεθών αυτών των ασφαλιών, τι θα σήμαινε αν ένα σημαντικό τμήμα αυτών των κινδύνων επαληθευόταν σε σχέση με εγκεκριμένε και αποδεκτέ ασφάλειες, σε σχέση για παράδειγμα με το ίδιο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο θα το ξεπερνούσαν. Ευχαριστώ. <clears throat> Καταρχάς, να επαναλάβω αυτό που ήδη είπα. Ακόμα και πριν ξεκινήσουν οι αναταράξεις που έχουμε εντοπίσει στις 9 Αυγούστου 2007 στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεχόμαστε ιδιωτικά έγγραφα και όχι μόνο πιο επίσημα των ε, κεντρικών ταμείων των Υπουργείων Οικονομικών και δεχόμασταν και σαν εγγυήσει και τα τραπεζικά αξιόγραφα όταν άλλοι δεν τα δεχόταν και δεχόμασταν και δάνεια. Άρα είχαμε ένα ευρύτερο πλαίσιο εγγύησεων. Διευρύνθηκε στο μη συμβατικό μέτρο. Εν συγκρίση με την έναρξη όμως, όχι πολύ. Προφανώς. Τι έγινε. Με τις αναταράξεις και την κρίση που ξέσπασε μετά το Σεπτέμβριο πέρσι, Ήθελαν οι τράπεζες να μας παρουσιάσουν αυτά τα ιδιωτικά έγγραφα αντί τα δημόσια χρεόγραφα που μας παρουσίαζαν πριν. Δίκιο έχετε. Ε, συμφωνώ. Η εκπνοή, η λήξη αυτών των εκτάκτων μέτρων απαιτεί κλιμακούμενη μεταβολή της συμπεριφορά των τραπεζών. Και αυτό ισχύει για αυτό που υπογραμμίσατε. Και ισχύει και για τη δυνατότητα που έχουν για να χρηματοδότηση για ένα χρόνο ή έξι μήνες. Στην αρχή της κρίσης, σταθερή κατάσταση, η μόνιμο μέτρο ήταν τρεις μήνες, όχι έξι μήνες, όχι ένας χρόνος. Αυτή είναι η έννοια της εξόδου, διεξόδου. Δεν είναι τώρα η στιγμή ε, εξόδου. Θα έρθει η στιγμή όμως. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή θα πρέπει να αναλυθούν αυτά που θέσατε. Δημοσιεύουμε όλα μας τα στοιχεία. Δεν θα σας κάνω να βαρεθείτε παραθέτοντας στοιχεία. Θα έλεγα όμως ότι το ερώτημά σας είναι πολύ καλά στοχευμένο είναι εύστοχο. Γιώργαν Κλούτ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μου δίνετε τον λόγο. Θα ήθελα και πάλι να επανέλθω στον Λόρδο Τέρνερ όπου έγινε αναφορά σχετικά και μια διαφορετική τοποθέτηση έκανε δημόσια που δίνει μια άλλη ματιά για τα αίτια της χρηματοοικονομικής κρίσης με πολύ επικριτικό τρόπο αναφέρθηκε σε σχέση με τα ε, τεκτενόμενα και ανέφερε επικρίσεις ε, συνολικά στις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα και είπε ότι είναι υπερβολικά φουσκωμένος ο χρηματοοικονομικός τομέας συνολικά. Αυτό μπορεί να είναι μια επίπτωση λανθασμένης αν θέλετε αναλογίας και επιμερισμού αναλογιών. Δική μου ερώτηση, πώς κρίνετε εσείς ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτό. Βλέπετε την δυνατότητα να επανέλθει στο κανονικό μέτρο των πραγμάτων ο χρηματοοικονομικός τομέας σε σχέση με την ε, υπερβολική, ας το πω έτσι, ε, εξόγκωσή του και σε σχέση με τις δυνατότητες για μια τέτοια αλλαγή ε, των χρηματοοικονομικών αγορών. Πώς το βλέπετε. Ο Λόρδος Τέρνερ είναι υπέρ ενός φόρου τόμπιν. Αυτό θα ήταν μια δυνατότητα για τον χρηματοοικονομικό τομέα να τον, να τον κρατήσουμε σε μικρότερες διαστάσεις, σε κάποιους τομείς. Τίθεται φυσικά το, ερώτημα, οι προϋποθέσεις ε, από το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο θα απορρεύσουν ή τι θα γίνει. Και στην ε, ε, σύνοδο των 20 κρατών στο Λονδίνο τον Απρίλιο, ο Κινέζος Υπουργό υπέβαλε μια πρόταση από πλευρά του να μην είναι το δολάριο το νόμισμα αναφοράς και να μην αντικατασταθεί με το ευρώ όπως λένε κάποιοι αλλά αν, αντί ενός κύριου νομίσματος να υπάρξει μια, ένα μείγμα αναφορών νομισματικό για την αντιμετώπιση της κρίσης. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. You have a lot of very, very Πολλά, πάρα πολύ σημαντικά σημεία τέθησαν να πω πώς ερμηνεύω εγώ τα όσα συνέβησαν. Είδαμε πόσο εύθραυστος ήταν ο παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός τομέας. Άρα πόσο εύθραυστη ήταν η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο εύθραυστη ήταν όλοι οι φορείς που είναι οι συνιστώσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να δεχο... ζούμε σε έναν τόσο εύθραυστο κόσμο. Έλλειψη αντοχής και αντίστασης είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Θεωρώ ότι όπως μια ασθένεια που είναι πολύ σκληρή και σοβαρή χρειάζονται πολυσχηδείς λύσεις και φάρμακα. Θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να βρούμε από αποδιοπομπαίους τράγους των παγκόσμιων δημοσιονομικών. Αν βρούμε αποδιοπομπαίο τράγο και πούμε η Τράπεζα Επενδύσεων, ε, οι φορείς βαθμονόμησης κλπ. φταίνε, τότε σώζονται οι άλλοι. Δεν εστιαζόμαστε στους άλλους. Τα πάντα πρέπει να αλλάξουν, τα πάντα, όλα πρέπει να διορθωθούν. Και χαίρομαι ιδιαίτερος διότι αυτό κάνουμε συμφωνούμε επί της μεθοδολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο αναδειωμένων οικονομιών και του βιομηχανικού κόσμου, του βιομηχανοποιημένου κόσμου και προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα πάντα. Και δεν θεωρώ ότι οποιοδήποτε κομματάκι δεν χρειάζεται σημαντική βελτίωση. Το όλο σύστημα ήταν εύθραυστο, το σύνολο ήταν εύθραυστο. Όσον αφορά το φόρο Τόμπιν, είμαι κατά τουλάχιστον αν πρόκειται περί του φόρου που είναι γνωστός ως φόρος Τόμπιν, περί τέτοιας φορολογήσεως, δεν θέλω να επεκταθώ, είμαι κατά όμως του φόρου Τόμπιν. Όσον αφορά το δολάριο, έχω να πω ότι επί του παρόντος είναι σημαντικότατο να μπορούμε σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας και παγκοσμίων ε, οικονομικών, δημοσιονομικών, έχουμε ένα ισχυρό δολάριο. Το δολάριο που θεωρείται ισχυρό από τις αρχές των ΗΠΑ, ως το θεωρούν οι αρχές της ΗΠΑ. Δηλαδή, ένα ισχυρό δολάριο είναι προς όφελος των ΗΠΑ, λένε οι Αμερικανοί και το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι αληθεύει και ότι αυτό που λένε οι Αμερικανοί για το πόσο σταθερό είναι το δολάριο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Τζέφρι Μπλουμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για το χρόνο σας κύριε Πρόεδρε. 35 χρόνια έχω περάσει σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υπό διάφορες ιδιότητες. Εγώ τα βλέπω από διαφορετική σκοπιά κάπως τα πράγματα οι περισσότεροι πολιτικοί δεν τα καταλαβαίνουν πολύ καλά τα οικονομικά θέματα. Ο, λέμε ότι ξεκινήσαμε από τους Lehman Brothers και κατηγορούνται όλες οι τράπεζες όπως η Solomon κλπ. Θα ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Εγώ πιστεύω ότι ξεκίνησαν τα γεγονότα από τους Αμερικανούς πολιτικούς οι οποίοι έφεραν τον ε, φόρο κοινοτικής επανεπένδυσης δεν αναφέρεται ότι ήταν τμήμα πολιτικών μεθοδεύσεων του χειρίστου είδους, το ενστερνήθηκαν οι τράπεζες, το χρησιμοποίησαν οι τράπεζες αυτό, κέρδισαν, στηρίχθηκαν τους πολιτικούς με χρήματα φορολογωμένων, από τους πολιτικούς που έκαναν τα λάθος, οι ρυθμιστικές αρχές έκαναν επανειλημμένα σφάλματα, ο Λόρδος Τέρνον αναφέρεται, και πήραν διάφορα στελέχη 10% αυξήσεις, μπόνους κλπ. και είχαμε τη μεγαλύτερη κατάρρευση τράπεζας στην ε, Ευρώπη. Μήπως θα έπρεπε Αυστραλία και Καναδάς να δούμε τι γίνεται εκεί. Δεν είχαν πρόβλημα. Οι Αυστραλιανές και οι Καναδικές τράπεζες έχουν άλλου είδους ρύθμιση και δεν αντιμετώπισαν προβλήματα ε, που δεν είναι τόσο περιοριστικό το πλαίσιο και κάποιος έπρεπε να υπερασπιστεί τον φορολογούμενο που τελικά έπρεπε να πληρώσει την ύφη. Όπως είπα, λέει ο Θεωρώ ότι τα παγκόσμια οικονομικά και δεν θα πρέπει να ξεχωρίζουμε κάποια κομμάτι όλα τα παγκόσμια η παγκόσμια οικονομία ήταν πάρα πολύ εύθραυστη ανώμαλα εύθραυστη έδειξε έλλειψη αντίστασης και οδηγηθήκαμε σε ελεύθερη πτώση της παγκόσμιας οικονομίας αυτό πρέπει να διορθωθεί βέβαια εντοπίζοντας το τι πρέπει να πράξουμε, είναι ξεκάθαρο ότι τεχνικά συστήματα τα οποία απεδείχθησαν τα πλέον ανθεκτικά θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικότατα. Διότι μπορούμε να μάθουμε πολλά μαθήματα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Επί παραδείγματι, βλέποντας τον Καναδά, βλέπω ότι η καναδική προσέγγιση όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Καναδά ε, ήταν ε, καλό, ήταν, αντιστάθηκε το καναδέζικο σύστημα. Δεν ξέρω να επενέσω τον Καναδά, αλλά πράγματι πρόκειται περί παραδείγματος που υπήρξε αντίσταση, άντεξε το σύστημα. Πέλτς. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Εντυπωσιάστηκα από αυτά τα οποία αναφέρατε στο ESRB. Ιδίω όπω ε, εξηγήσατε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εσεί, αλλά και ε, ο Αντιπρόεδρος ε, εμπλέκεστε στο Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με αυτό το εγχείρημα. Τις τελευταίες εβδομάδες έμαθα ότι και προειδοποιήσεις και συστάσεις μπορεί να διατυπώνεται. Ερώτησή μου, θα μπορούσε ίσως να καταλήξετε σε μια κατάσταση που θα πρέπει να δικαιολογήσετε κάποια πράγματα όταν ε, είδους, ε, τέτοιου είδους συστάσεις ή προειδοποιήσεις ε, δεν επαληθεύονται από πλευρά σας και θα πρέπει να δικαιολογείται τις πράξεις. Και τι γίνεται σε σχέση με τον πριτανεύοντα στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μια ανεξάρτητη νομισματική πολιτική που πρέπει να διασφαλίζεται. Συγκεκριμένη ερώτηση, μήπως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εδώ όσον, σας, όσον αφορά εσάς. Δεύτερη ερώτηση που έχω. Πριν έρθω στην Ευρωβουλή, ο ίδιος 15 χρόνια ήμουν, είχα δραστηριοποιηθεί στο χρηματοοικονομικό τομέα, στο πιστοτικό τομέα. Είχαμε την συζήτηση πανευρωπαϊκά τι είναι τα συστημικά και τι ε, είναι τα συστημικά ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κανεί δεν μπόρεσε να μου απαντήσει αυτό το ερώτημα. Ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να βοηθήσει στην απάντηση του ερωτήματο. Η τρίτη μου ερώτηση, μια και πρέπει να ολοκληρώσω, αφορά τα κρατικά ε, ταμεία, τα ταμεία αυτά τα αποθεματικά εκτός ζώνης ευρώ. Αυτά τον τελευταίο 1,5 χρόνο συνεισέφεραν για τη σταθερότητα της διεθνούς οικονομικής επιστοτικής αγοράς. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ήδη ανέφερα, θα απαρτίζεται από διάφορους συμμετέχοντες αυτός ο φορέας, το ECRB. Θα έρχονται και παρατηρητές όπου τη χρειάζεται, εκπροσωπώντας τις διάφορες ε, εποπτικές αρχές. Σύγκρουση συμφερόντων, σίγουρα όχι, διότι η ίδια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη συνθήκη του Μάστριχτ, είναι το κέντρο για την νομισματική πολιτική, όπως είπα στην εισαγωγή μου, και η σύσταση που θα κάνουμε όσον αφορά την μακροεποπτεία οι συστάσεις που θα κάνουμε ίσως να μην διαφέρουν κατά πολύ από αυτά που λέμε εμείς όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, την ανάγκη διαθροτικών μεταρρυθμίσεων. Κάνουμε συστάσεις στον τομέα. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά ίσως να σχηματίζεται μια ιδέα πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα πράγματα. Και δεν θα έχουμε εκτελεστική αρχή δεν θα έχουμε μάλλον εκτελεστική εξουσία και κύρος. Θα είναι συστάσεις απλές που θα κάνουμε. Όταν συζητούμε την Επιτροπή σας θα είμαστε υπεύθυνοι να αξιολογούμε τις συστάσεις. Πολύ συχνά συζητούμε τα θέματα των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων, εν είναι ή λάθος. Στους διάφορους τομείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πράγματα. Και είναι ένα κομμάτι των καθηκόντων μας όσον αφορά τα συστημικά χρηματοπιστωτικά χρηματοστηρικούς φορείς. Εκεί δυστυχώς είχαμε μεγάλα παραδείγματα αυτών. Όταν κυβερνήσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού αποφάσισαν να, προσπα... να δοκιμάσουν να αποφύγουν καταστροφικά συμβάντα Σωστή ήταν η κρίση τους πιστεύω. Σε μια περίπτωση είδαμε ότι ένα γεγονός μπορούσε να δημιουργήσει σε όλο τον κόσμο συγχρονισμένες αποφάσεις σε όλο τον κόσμο. Βλέπαμε λοιπόν ότι αυτό η συστημική πτυχή, το συστημικό γεγονός ήταν κάτι που ίσχυε, ήταν θέμα κρίσεως βέβαια. Δεν ξέρω τι να πω όσον αφορά τα κρατικά τάμια, τα κυβερνητικά τάμια, τους κυβερνητικούς πόρους, αν αυτό ήταν το ερώτημά σας. Εξακολουθούν να παίζουν το ρόλο τους, σε, αυτή την, σε αυτό το στάδιο όμως δεν μπορώ να κρίνω. Αλφρέντο Παλώνε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Τρισέ, έχω ερωτήσεις όσον αφορά τους ε, κανόνες. Διότι βλέπω όσον αφορά τις τρεις αρχές. Μου ήρθε στο μυαλό πως οικοδομήθηκε η διαδικασία που αφορούσε το ενιαίο νόμισμα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω μιας μεγάλης διαδικασίας δημοκρατικής με μεγάλη αυτονομία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ερώτημα λοιπόν. Διάβαζα τον κανονισμό και μου δημιουργήθηκε σύγχυση λόγω ενός κειμένου. Λέει ότι εκ των πραγμάτων εξαιρείται να μπορούμε να βρεθούμε στην κατάσταση που το βασικό όργανο του Ευρωπαϊκού Συστηματικού, Συστημικού Συμβουλίου η Διευθύνουσα Επιτροπή δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι κάτι που με μπέρδεψε. Βλέπω τις τρεις αρχές μετά που αναφέρονται. Όπως συνέβη και σε εσά δεν εκλέγονται άμεσα τις κυβερνήσεις και από τα κοινοβούλια, αλλά από τα μέλη του Συμβουλίου των Εποπτικών Αρχών. Λοιπόν, κύριε Δικητά, κύριε Τρισέ, δεν πρέπει να εγγυηθούμε δύο πράγματα. Όσον αφορά τη μάκρο και μικρο εποπτεία για τη συνετή διαχείριση που θέλουμε να ενισχυθεί, να ενισχύσουμε τελικά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι να την αποδυναμώσουμε. Γιατί θυμηθείτε και θέμα κύρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και πρέπει να τεθεί στο θέμα σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων και όχι μόνο σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων των διαφόρων εποπτικών φορέων που ε, κινούνται στις διάφορες χώρες μας. Δηλαδή να τεθεί πιο πολύ το θέμα σε επίπεδο κυβερνήσεων, πιο κοντά στο, στους λαούς. Απάντηση, αν κατάλαβα καλά. ασχολείστε με την πρόταση που γίνεται σε επίπεδο μικροεποπτείας. Το επεξεργαζόμαστε το ζήτημα. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν εμπλεκόμαστε άμεσα, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουμε τι γίνεται στα πλαίσια της κανονικής διαβούλευσης. Προσπαθούμε να μελετήσουμε τα προτινόμενα για την μικροεποπτεία. Ξέρουμε πολύ καλύτερα τον μακροοικονομικό φορέα της διαχείρισης. Γιατί πολύ συχνά έχουμε συζητήσει σε αυτό το επίπεδο, έχουμε εμπλακεί σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός όσον αφορά τα σχόλιά σας που αφορούσαν την μικροεποπτεία και τις σχετικές αρχές. Ελπίζω να με συγχωρέσετε γι' αυτό. Θα δούμε ποια θα είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα πρέπει να αποφανθεί. Κάποια στιγμή είπατε νομίζω ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν συμμετέχει σε κάτι. Τι, τι εννοούσατε, τι λέτε. Εκτός μικροφώνου ο διάλογος του κυρίου Τρισέ με τον Ιταλό. Θα μπορούσε να μην συμμετέχει, λέει ο κανονισμός. Θα μπορούσε να μην συμμετέχει. Απάντηση. Επιστρέφεται στην, στις αρχές μικροεποπτείας, εποπτείας σε μικροοικονομικό επίπεδο. Κάτι προτείνεται από την ε, ομάδα Λαροζιέρ. Ε, Οι περισσότεροι βουλευτές είχαν αντίθετη άποψη. Μας έλεγαν ότι πρέπει να αναμειχθείτε στην εποπτεία σε μικροοικονομικό επίπεδο. Δεν ήταν αυτό πρόθεση της ομάδας Λαροζιέρ ούτε, ούτε προθέσει του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως θα αποφασίσετε εσείς. Αλλά για μένα ήδη είναι η λιμένη απόφαση αυτή. Αποφασίστε και προκαιρού. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και να σας απαντήσουμε εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου. Διότι μιλάμε πάντα για μια διαδικασία διαβούλευσης. Επόμενος. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ξεκινώ αμέσω με την τελευταία σας διαπίστωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Οδηγία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είπε με σαφήνεια ότι <clears throat> στην επιτήρηση θέλουμε ένα βήμα ολοκλήρωση που θέλουμε να γίνει και θέλουμε ενισχυμένα να εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμένα δεν μου επαρκούν αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται επί τραπέζης ως προτάσεις. Ιδιαίτερα υπό το πρίσμα αυτού που αναφέρατε, ότι δηλαδή έχουμε μία παγκοσμιοποιημένη ε, χρηματοοικονομική συναλλαγή αλλά δεν έχουμε ούτε καν ευρωπαϊκή επιτήρηση. Δεν έχουμε φτάσει αρκετά μακριά λοιπόν όσον αφορά την, την επιτήρηση. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε μαζί μου. Το άλλο σημείο και εδώ σε σχέση με το ερώτημα, ποιο κόστος προκαλεί η ε, διαδικασία αυτή όσον αφορά το θέμα των ιδίων κεφαλαίων και όσον αφορά τους κανόνες χρηματοδότησης. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα, διότι το φθινόπωρο πρέπει να συζητηθεί αυτό. Το τρίτο σημείο ως παρατήρηση είναι, είπατε ότι το πρόβλημα έγκυται στην διάθρωση, στη δομή και όχι στα επιμέρους προϊόντα ή στους επιμέρους φορείς. Το συμμερίζομαι αυτό τα διαθωτικά προβλήματα θα μπορούσατε να τα αναφέρετε υπό αυτό το πρίσμα ότι πρέπει να τα αποφύγουμε. Και τελευταία ερώτηση πληθωρισμός και λόγω χρεών και δυνατότητα exit στρατηγικής ε, ε, διεξόδου και βλέπουμε εδώ σε σχέση με το εύκολο χρήμα πώς το βλέπετε σε σχέση με το όριο των 2, του 2% ποιο ρόλο διαδραματίζει η πολιτική αντιμετώπιση χρεών για τη στρατηγική διεξόδου exit από την κρίση για σας Thank Ευχαριστώ Όσον αφορά το πρώτο σχόλιο, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαι ικανοποιημένος γι' αυτό, αυτό που αποφασίστηκε σε επίπεδο G20 που συμπεριλαμβάνονται και, και σε άλλα βήματα που συμπεριλαμβάνονται και χώρες του βιομηχανικού κόσμου και του αναπτυσσόμενου κόσμου χρησιμοποιούμε τις ίδιες αρχές και πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ίδιες αρχές. Εάν θέλουμε να είναι πιο ανθεκτικό το σύστημα, χρειάζεται να είναι ισότιμοι οι όροι, οι ίδιες αρχές να ισχύουν παντού. Αυτή ήταν η θεωρία της παλιάς Επιτροπής της Βασιλείας. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της φοβερής κρίσεως της δεκαετίας του 80, του Sovereign Risk. πάντα υπήρχε αυτή η ανάγκη να, υπάρχει, να υπάρχουν αρχές και κανόνες συνετής διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Εφαρμόζονται σωστά ή όχι. Κρίνετε εσείς. Ήταν σαφές ότι σημαντικές βελτιώσεις έπρεπε να γίνουν για τη σωστή εφαρμογή των ίδιων αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ζητάμε από έναν φορέα να είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή αυτών των κανόνων και η έννοια αυτή βασίζεται σε εφαρμογή από συστάδα αρχών, σε παγκόσμιο επίπεδο σίγουρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω πολύ καλά τη θέση σας. Την καταστήσατε σαφέστατη. Και εδώ. Εγώ θα έλεγα είναι πολύ καλή ιδέα να υπάρχει μία αρχή στην Ευρώπη που θα σκεί αυτή την μικροεποπτεία. Αλλά δεν προτάθηκε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι απίθανο να υπάρξει η δυνατότητα να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των διαφορών χωρών σε αυτή τη φάση. Ξέρω ότι σας λυπεί αυτό. Αλλά σε αυτή τη φάση τίνω να πιστεύω ότι είναι γεγονός. Αλλά είναι έτσι σημαντικότερο τότε να είμαστε σίγουροι ότι οι ίδιες αρχές, στην περίπτωση της Ευρώπης, η ίδια οδηγία στην περίπτωση της Ευρώπης εφαρμόζεται δίκαια, ακριβώς πανομοιότυπα σε κάθε χώρα. Όσον αφορά την στρατηγική εξόδου, μου λέτε ότι δεν χρειάζεται μόνο να ξεφύγεις, να βγεις από τα μη κανονικά μέτρα, αλλά χρειάζεται να σκίσεις τη δική σου νομισματική πολιτική και να αποφασίσεις για τα επιτόκια σου. Πάντα αυτό το έλεγα, ότι αυτό εξυπακούεται. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ούτω ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να σας λέμε σε εσά και στους συμπολίτε μας ότι εξασφαλίζουμε μέσω μακροπρόθεσμα σταθερότητα τιμών και στο τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να αποτιμήσουμε τα πεπραγμένα από όταν δημιουργήθηκε το ευρώ για, την, για τα πρώτα 11 χρόνια. Όταν κάνουμε αυτή την αποτίμηση θα δείτε ότι ανταποκριθήκαμε στην εντολή που μας δώσατε, την πρωταρχική εντολή που μας δώσατε εσείς, οι δημοκρατίες της Ευρώπης. Και οι συνάδελφοί μου και εγώ είμαι υπερήφανοι γι' αυτό. Αλλά το ότι είμαστε αξιόπιστοι στο μέλλον, για το μέλλον, Γι' αυτό, για να είμαστε αξιόπιστοι στο μέλλον, γι' αυτό στα επιτόκια, τα μέσο και μακροπρόθεσμα έχουμε την έννοια της σταθερότητας των τιμών. Κάτω από δύο, κοντά στο δύο, κάτι που είναι αξιόπιστο για όλους. Και τους επενδυτές και τους αποταμιευτές και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ, ο Έντουαρντ. Όπως και συνάδελφοι θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω ε, για την, το ότι ήσασταν διαθέσιμος και απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Ε, ε, αλλά θα πρέπει η δεξιά να γνωρίσει τι κάνει η αριστερά. Χείρα. Όσον αφορά τη μία πλευρά ήσασταν σαφείς για την στρατηγική εξόδου δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να εξέλθουμε αλλά όσον αφορά τη φορολογία στην Ευρωζώνη νομίζω ότι είναι πιο ασαφής η κατάσταση. Οπότε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μειώσουμε ε, τα, ούτε να αυξήσουμε ούτε να μειώσουμε τα οικονομικά κίνητρα αλλά συσφίγγει τις διαδικασίες δυσιονομικών ελλημάτων που είναι ένας τρόπος λογιστικής πιέσεως. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να περιμένει για μια χώρα να δείξει κάποια ανάκαμψη προτού η χώρα αυτή να μπορέσει να μειώσει το έλλειμμά της Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνούμε και στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, δύσκολη λειτουργία της για να ε, ε, εφαρμόσει το σύμφωνο σταθερότητος είναι και ένα θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν οι επενδυτές και οι αγορές δεν έχουν το συνέστημα ότι η δημοσιονομική κατάσταση είναι υποέλεγχο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, μία ανάκαμψη. Οπότε θα ήθελα απλώς να σας πω ότι το μήνυμα το οποίο δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνούμε πλήρως με αυτό σχετικά με το επίπεδο ε, είναι η αρχή της της ανακάμψεως για τη φορολογική πολιτική ε, θα είναι μόλις ξεκινήσει η ανάκαμψη με μία αύξηση των φορολογικών συντελεστών το 2011. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμεί συμφωνούμε πλήρω. Βέβαια, ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες όσον αφορά ε, το, ε, τα χρέη τους σε σχέση με ε, το ΑΕΠ και το μέγεθος των ελλημάτων και όλα αυτά καλύπτονται από την αγορά, από τους αποταμιευτές και από τους πολίτες που χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Είναι δηλαδή πολύ βασικές παράμετροι, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει ε, ε, ασυμβίβαστος στις απόψεις μου. Δηλαδή πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να επανέλθουμε σε ένα αίσιο κλίμα και να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη διότι η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι η οποία οδήγησε στην τωρινή κρίση. Ευχαριστώ. Κύριε Τρισέ, η πρόσφατη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και οι ελπίδες ε, για ε, μία ανάκαμψη είναι μία πηγή ε, αισιοδοξία για τις χώρες που θα προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη. Αλλά είπατε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν περιμένουν να υπάρξει μία αύξηση πέραν του 3% και για τα νέα κράτη-μέλη ε, η ανάγκη ισοσκελίσεως των ε, ισολογισμών τους ε, είναι σε σύγκρουση με τα χαρακτηριστικά του Μάστριχτ και ε, με τις αρχές του Μάστριχτ και ε, υπάρχει το θέμα της ασυμμετρικής ε, ρευστότητος όπως και άλλα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και το ερώτημά μου είναι δεδομένων όλων αυτών τι άλλα μέτρα πιστεύετε ότι χρειάζονται για να μπορέσουν τα νέα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη και για να παραλληλήσω με τα προηγούμενα σχόλιά σας ποιο είναι το φάρμακο που προτείνεται στην παρούσα κατάσταση. Ευχαριστώ. Θα σας έλεγα ότι η προσχώρηση στην Ευρωζώνη είναι θέμα στρατηγικής θέλησης, πολιτικής θέλησης με ευγενή διατύπωση δηλαδή πολυκομματικής θέλησης και όταν υπάρξει μία πολυκομματική συνένεση δεν είναι, δεν είναι περίεργο διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, προσπαθεί να καλύψει όλες τις ευαισθησίες. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Δεύτερον υπάρχουν τα κριτήρια και τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ε, για να αναθεωρήσουμε τα κριτήρια στην Ευρωζώνη και ε, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να συνεργαστούν για να συνεννοηθούμε Κάθε τρίμηνο έχουμε στοιχεία, έχουμε μια συνεχή επαφή, τεχνική βοήθεια κάθε είδους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός των 27 ε, χωρών και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά και η εποπτική, το Εποπτικό Συμβούλιο που προτείνουμε θα συμβάλλει σε αυτή την συνεννόηση. Βέβαια, δικιά μας ευθύνη είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την τάξη στην Ευρωζώνη γιατί η Ευρωζώνη είναι βασικό στοιχείο και το γεγονός ότι είμαστε στα πόδια μας είναι πολύ βασικό. Θα πρέπει όμως όλοι να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε αυτή την καλή λειτουργία, σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε 25 χώρες στο ευρώ. Ευχαριστώ κύριε Τρισέ. Ελπίζω να έχουμε 25 χώρες, ενδέχεται όμως να υπάρχει μία λιγότερη. Προσπαθώ να καταλάβω τις επιπτώσεις των προτάσεων των επιτροπών, της Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα. Και δεν είναι πολύ σαφές, μπορείτε ίσως να με βοηθήσετε κύριε Τρισέ. Ε, το ESRB δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Ε, είναι μια σύσταση. Η σύσταση όμως που απευθύνεται στα τα κράτη-μέλη και στους διάφορες οργανώσεις ε, δεν ε, βρουν τα απόκριση σημαίνει ότι το κύρος της ESRB θα μειωθεί Συμφωνώ μαζί σας ότι το ευρώ και η ευρωζώνη είναι μία άγκυρα ε, κατά την κρίση όχι μόνο για τις χώρες του ευρώ. Επίσης όσον αφορά τη συμμετοχή της ε, ESRB θα μπορούσατε να επιλέξετε ε, διοικητές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δεν θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ε, προεδρεύει στην ESRB, στο ε, Εποπτικό Συμβούλιο. Και τέλος μία τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι η Ευρώπη ενώθηκε κατά αυτή την κρίση. Ίσως όμως διαιρέθηκε και περισσότερο. Έχουμε ε, τις χώρες της ε, Ευρώπης από τη μια μεριά και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε πιο ευέλικτη ε, ερμηνεία των κριτηρίων όπως προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ευχαριστώ. Σχετικά με το πρώτο θέμα που είναι πολύ βασικό όπως έχει το κείμενο τώρα, είναι θέμα κρίσεως. Εάν δηλαδή η σύσταση της ESRB ε, δημοσιοποιηθεί ή όχι. Είναι, είπατε ένα θέμα κρίσης, αλλά και η δημοσιοποίηση ε, είναι λεπτό θέμα και ελπίζω ότι η σωστή κρίση θα μπορέσει να πρεσβεύσει διότι αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς θεωρείτε ότι ε, αν ε, υπάρχει μία σύσταση η οποία βασίζεται στη ε, τη συμμόρφωση και στις εξηγήσεις η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Βέβαια εάν προχωρήσετε στη συλλογιστική αυτή δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή αν πιστεύετε ότι και οι συστάσεις χωρίς ε, αλλαγή της αρχής θα είναι αντιπαραγωγικές εγώ θα ήθελα να σας απαντήσω ότι μπορεί ε, να είναι δημόσια και να είναι πιο αποτελεσματική αν δεν γίνει ε, δημόσια, δεν κοινοποιηθεί δηλαδή η κατάρτισή της. Όσον αφορά τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ESRB, θα είναι ε, το Κεντρικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Οι συνάδελφοί μου και εγώ δηλαδή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω καλύτερα. Πρέπει να είμαστε εκεί. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να προσπαθήσει να αλλάξει την πρόταση. Νομίζω όμως ότι η πρόταση αυτή είναι σωστή για να σας πω την αλήθεια. Διότι έχετε τους 27 στο Γενικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οπότε ε, θα είναι προφανές ότι είμαστε στο επίπεδο των 27 και όχι ε, μόνο σε ε, μία περιοχή. Νομίζω ότι αυτή ήταν η ιδέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όταν το σκέφτηκε. Θα σας πω επίσης ότι δεν νομίζω ότι θα κάνουμε καλό στην Ευρώπη εάν αλλάξουμε τα κριτήρια. Εν πάση περιπτώσει, η είσοδος στην, ε, ε, στη ζώνη του ευρώ δεν είναι κάτι το οποίο ε, θα σας, θα σας θα σας προφυλάξει από δύσκολες μέρες είναι μία απόφαση που πρέπει να πάρετε και θα συμμετέχετε στα τεκτενόμενα οπότε ε, νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε τα κριτήρια και είναι καλή ιδέα αυτή για να είμαι Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Τεράστια ευχαρίστηση να μπορεί κανείς να σας ακούσει και σε σχέση με την ερώτηση που απαντήσατε. Η άλλη ερώτηση είναι τα κριτήρια σύγκλησης. Πιστεύετε ότι πρέπει να τηρηθούν. Απαντήσατε σχετικά και πιστεύω ότι όχι μόνο στα νέα κράτη-μέλη βέβαια, διότι ερωτούν οι πολίτες για τον ορθολογισμό ή τα άλλα κράτη-μέλη. Τι γίνεται με τα κριτήρια αυτά. Κάποιοι λένε ότι αφορούν τους εκτός ε, της ζώνης ευρώ κιόλα. Η ερώτησή μου όμως είναι η εξής. Στις χώρες εκείνες που έχουν υποβάλει αίτηση να ενταθούν στην Ευρωζώνη, πολύ συχνά αναφέρεται ότι ουσιαστικά είναι μια πρόκληση που περιορίζεται στις ίδιες αυτές τις χώρες. Δεν υπάρχει μια γενική πολιτική δηλαδή συνολικά που θα ε, βοηθούσε τις χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Η ικανότητα να ενταχθούν στην Ευρωζώνη και το να είναι κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ε, κάποια κράτη βοηθά σίγουρα θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη διεύρυνση της ζώνης ευρώ. Αν ναι, τότε τι θα έκανε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τι θα έλεγε για αυτή τη στρατηγική. Ποια θα ήταν η δική σας άποψη δηλαδή για μια τέτοια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ευχαριστώ. Διαπραγματεύτηκα τη συνθήκη του Μάστριχτ με τους συναδέλφους υπουργό εσωτερικών, διάφορους φορείς και τον πρόεδρο της Γερμανίας, Καγελάριο, με τον Υπουργό Εξωτερικών, συζητήσαμε το θέμα και θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει η Ευρωζώνη με έξι χώρες, έξι-επτά χώρες, ούτως ώστε να έχουμε την κρίσιμη μάζα. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τότε θεωρούσαν ότι ίσως να είναι δυνατόν μόνο δύο χώρες να ξεκινήσουν με το ευρώ είπαν εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ξεκινήσουμε πριν το έτος 2000, πρώτη πρώτου 99. Αποφασίστηκε στο Μάστριχτ, ακόμα και αν συμπεριλαμβάνονται μόνο δύο χώρες. Ξεκινήσαμε 11. Πρώτη πρώτου 99, 11 χώρες. Φανταστικό. Και απόδειξη ότι η έννοια της Ευρωζώνης ήταν ε, κάτι που κάλυπτε πολύ μεγαλύτερο αριθμό χωρών από αυτό που προβλεπόταν τη στιγμή των, ε, την ώρα των διαπραγματεύσεων. Τότε πολύ γρήγορα ήμασταν 12, σήμερα είμαστε 16 συμπεριλαμβανομένων δύο πρώην κομμουνιστικών χωρών στην Ευρωζώνη, στην καρδιά της Ευρωζώνης. Οπότε δεν είναι κλειστό κατάστημα αν θέλετε, δεν πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Κάθε χώρα αποφάσισε να μπει. Όχι διότι εφαρμοζόταν μια στατηγική και μόνο, αλλά διότι θεώρησαν οι χώρες αυτές ότι ήταν έτοιμες, θεώρησαν ότι έπρεπε να μοιραστούν το κοινό πεπρωμένο, ήταν πολλές ευαισθησίες που εκφραζόταν σε αυτό το συνέστημα και υπήρχαν και κριτήρια. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. 16 χώρες και ξεκινήσαμε με 11. Είναι μεγάλη αύξηση αυτή. Μιλάμε για ένα ιστορικό φαινόμενο. Με τα μάτια του ιστορικού, αν τα δει κανεί, αν δει κανεί αυτή την ιστορική διαδικασία, είναι αξιοσημείωτο γεγονό και θα συνεχίσουμε τη διεύρυνση. Πρέπει να συνεχίσουμε τη διεύρυνση επί τη βάση της σωστής προετοιμασίας, της απαραίτητης σύγκλησης. Ορίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε την Ευρωζώνη και βρισκόμαστε εμείς εκτός Ευρωζώνης, είμαστε όμως μέρος του υπολείπου και δυστυχώς η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε, που χρειάζεται την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει τα πλήγματα τις περισσότερες φορές είχε ακολουθηθεί λανθασμένη πολιτική, νομισματική και οικονομική πολιτική. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό και αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα τα προβλήματα. Βρισκόμαστε σε μια κρίση ακόμα. Οι τράπεζες δεν είναι πρόθυμες να διαθέσουν ε, δάνεια, πιστώσεις και υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ανάκαμψη και βρισκόμαστε μπροστά και σε μια ας το πω έτσι ταραχή θα πρέπει εδώ να δούμε το θέμα της διαχείρισης της κρίσης. Όπως προανέφερα, σε, προανφέρθηκε σε εσάς κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασής μας, ουσιαστικά η αρχή της ίσης ε, μεταχείρισης και ίσης ε, αντιμετώπισης δεν ήταν, δεν έγινε σεβαστή στην διαχείριση και αντιμετώπιση της κρίσης. Τον Οκτώβριο η Εθνική ζήτησε η ε, ε, τράπεζά μας ε, και δεν δόθηκε έγκριση. Στη Σουηδία, στην Δανία το swap επετράπει όμως. Βλέπουμε ότι σε άλλους δεν επετράπει. Αυτό τι δείχνει. Αυτό δείχνει δεν υπάρχει ίση μεταχείριση για τα μέλη εντός και εκτός της Ευρωζώνης. Ακόμα και για τα μέλη εκτός Ευρωζώνης πάλι αυτά δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα μεταξύ τους. Θα ήθελα να ζητήσω όταν θα θεσπιστεί το ESRB ερώτησή μου σημαντικό θα είναι σίγουρα για τα θέματα των Ευρωπαϊκών κρατών να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν σαν ένα τμήμα της πολιτικής αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων και βλέπουμε εδώ σε σχέση με την ε, Ουγγαρία έχουμε μεγάλα προβλήματα. Θέλω να ρωτήσω, έχει κάποια πρωτοβουλία που έχει υπόψη της να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ρωτήσατε. Το τελευταίο ερώτημα αφορούσε το ESRB. Ε, την Επιτροπή του Συστημικού Κινδύνου. Το τελευταίο σημείο θα ήθελα να καταλάβω. Κοιτάξτε, έχω ένα αίτημα και ένα ερώτημα. Όταν δημιουργηθεί αυτή η Επιτροπή του Συστημικού Κινδύνου, η e τότε η αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα, διότι έχουμε πικρές εμπειρίες ε, από το παρελθόν, όπως σας ανέφερα. Ήθελα λοιπόν να υποβάλω το αίτημα τα προβλήματα της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης να αντιμετωπιστούν υπό την ίδια αιγίδα και συγκεκριμένα όσον αφορά την Ουγγαρία έχουμε πολλούς δανειολήπτες που χρεοκόπησαν. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάποιες πρωτοβουλίες για να εξαλείψει αυτού του ίδιου τον κίνδυνο. Απάντηση. Να σας πω ότι πρώτα απ' όλα όταν χρησιμοποίησαμε αυτά τα έκτακτα μέτρα στην Ευρωζώνη ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της Ευρωζώνης στο ευρωσύστημα αυτό είπαμε στις τράπεζες μας ότι και στα παραρτήματά τους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ότι θα έπρεπε να εξακολουθούν να παρέχουν ρευστό στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Ήταν σαφέστατο το μήνυμα, σαν κρίσταλο. Και θεωρώ ότι ίσως να μην ήταν τόσο ορατό το μέτρο αυτό, αλλά ήταν ένας τρόπος να βοηθηθεί η χώρα σας και άλλες χώρες. Να πω ότι είχαμε και διμερή συμφωνία ρέπο με την Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας προς διευκόλυνση της ε, καταστάσεως που ήταν πολύ δύσκολη. Το ESRB είναι ένας θεσμός των 27, σωστά το είπατε, και θα πρέπει να αποφασίσουμε όσον αφορά τους κινδύνους για τις 27 χώρες. Ποια είναι η ιδέα να εξεταστεί το θέμα των δανείων σε ξένο νόμισμα που είναι ένα από τα προβλήματα που θέσατε και είναι τυπικά ένα θέμα που θα μπορούσε να εξεταστεί στο επίπεδο αυτής ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ε, επίπεδο 27. Ο Σόραν Τάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της ε, μου δίνει ιδιαίτερη χαρά να μπορώ να σας προσφωνήσω σήμερα εδώ. Συμφωνώ με τη δήλωσή σας ότι έκτακτοι καιροί απαιτούν έκτακτα ξεχωριστά μέτρα. Η απόφασή σας για διευρυμένη δανειακή υποστήριξη είναι κάτι που χαιρετίζουμε. Το ίδιο επίσης και η στρατηγική εξόδου από την κρίση. Όμως παραμένουν σαφή τα ε, γεγονότα. Τα επιτόκια του ευρώ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Τον Ιούνιο η Ευρωζώνη είχε αποπληθωρισμό που αντιμετώπισε για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τον Αύγουστο το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού ήταν ήδη 0,7%. Οι τράπεζες δίνουν ισχυρά αρνητικά μηνύματα προς τους δανειολήπτες η δανειοληπτική πίστη και η εμπιστοσύνη είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το να κρατηθούν τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα θα μπορούσε να είναι μεγάλη απειλή. Να θυμηθούμε την κρίση που πέρασε η Ιαπωνία την δεκαετία του 90 και σε σχέση με τα επιτόκια τον ρόλο που διαδραμάτισαν για την ανάκαμψη στην Ιαπωνία. Θα ήθελα λοιπόν μια σαφή απάντηση από πλευρά σας για τον κίνδυνο μιας αρχής σπυροειδούς εξέλιξης στασιμοπληθωρισμού ή αποπληθωρισμού στην ζώνη ευρώ, στην ευρωζώνη. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι η απουσία εμπιστοσύνη είναι ένα από τα κυριότερα εμπόδια για την ανάκαμψη της οικονομίας. Θα έπρεπε να έχουμε συνειδητοποιήσει το γεγονός από την άλλη πλευρά ότι όλο και χαμηλότερα επίπεδα φτάνει αυτή η σε εξέλιξη απουσίας εμπιστοσύνη, Υποστηρίζεται την άποψη ότι οι τράπεζες που βοηθήθηκαν με χρήματα των, των φορολογουμένων θα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα να βοηθήσουν τους ε, δανειολήπτες, τους ε, πολίτες. Πώς θα πρέπει, πώς θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε τι τράπεζε να, το κάνουν αυτό και ποιε ιδέε έχετε για να αναλυφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το φαινόμενο του τουρισμού. Είχαμε προβλέψει ότι θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού, ότι θα είμαστε σε αρνητικό πρόσημο για μια περίοδο και θα επανέλθουμε σε θετικό. Και όλοι το κατάλαβαν αυτό, η αγορά, οι παρατηρητές, οι διάφοροι φορείς που συμμετέχουν στο σύστημα και θα κάνουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Όλα αυτά οφείλονται στα βασικά αίτια. Δεν υπήρξε η υλοποίηση του αποπληθωριστικού κινδύνου στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο αυτό και στα μάτια των παρατηρητών. Όσον αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εμπιστοσύνη είναι αυτό που εξατμίστηκε τις 15 Σεπτεμβρίου πέρσι και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, σε όλους τις συνιστώσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πώς προσπαθούμε να το κάνουμε. Καλά μας τα είπατε. Προσπαθώντας να είμαστε τολμηροί όποτε αυτό χρειάζεται. Να χρησιμοποιούμε και έκτακτα μέτρα όταν χρειάζεται. Μη συμβατικά. Να είναι ηλίου φαϊνότερο ότι ποτέ μα ποτέ δεν δεχόμαστε να αποκλίνουμε από τον πρωταρχικό μας στόχο. Μέσω μακροπρόθεσμα δηλαδή να διατηρήσουμε τη σταθερότητα τιμών. Θέμα εμπιστοσύνη είναι. Διότι και οι προσδοκίε όσον αφορά τον πληθωρισμό ταιριάζουν με την στρατηγική μας για τη σταθερότητα τιμών μέσω μακροπρόθεσμα αλλά επί του παρόντος με πολύ χαμηλό πληθωρισμό για την προβολέ μας. Επιβεβαιώνουμε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το μήνυμα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο. Τελευταίο ερώτημα. Ο κ. Μπόκρος, έχουμε άλλα πέντε λεπτά διερμηνία. Δεν χρειάζομαι διερμηνία. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναπερφερθώ στο θέμα και θέλω να θίξω τα κριτήρια του Μάστριχτ. Σαφώς μας τα είπατε κύριε Κτρισέ ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση στα κριτήρια προσχώρησης και πρέπει να έχουν επίγνωση τα κράτη-μέλη. Το θέμα τίθεται κατά πόσο για τη συνοχή της Ευρωζώνης τι κάνουν αυτά τα κριτήρια. Κάποιοι λένε ότι η κρίση ίσως άλλαξε την οτροπία μας. Όσον αφορά την υφή των κριτηρίων του Μάστριχτ. Κάποιοι λέγουν ότι χρειαζόμαστε κριτήρια για, τους, για τα τρέχοντα έξοδα. Διότι αν έχει διπλό χρέος και έλλειμμα μια χώρα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πιο ευάλωτη από ότι αν έχει φορολογικό έλλειμμα. Άλλοι λένε ότι πρέπει να εξαλείψουμε το φορολογικό κριτήριο και αυτό. Διότι οι περισσότερες χώρες σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να ανταποκριθούν και στο προβλεπτό μέλλον δεν θα μπορέσουν. Τι σκέφτεστε εσείς. Δεν ζητώ από το διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μου απαντήσει, αλλά σαν θεωρητικός των οικονομικών θεμάτων, νομισματικών θεμάτων, πώς θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα αυτό για να αυξήσετε τη συνοχή της Ευρωζώνης. Απάντηση. Δεν μπορώ να διαχωρίσω τις ιδιότητες. Δεν μπορώ να χωριστώ στα δύο, λέει ο κ. Τρίσε. Να σας πω το εξή. Όταν λέω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τηρούμε τα κριτήρια, λέω ότι επαναλαμβάνουμε μόνο αυτά που λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτά που από ό,τι γνωρίζω λένε οι περισσότερες χώρες που δεν θα ήθελαν να ισχυριστούν ότι προσχωρούν εκμεταλλευόμενες μία ε, ασυνήθιστη κατάσταση και ότι δεν έχει επιτευχθεί η απαραίτητη σύγκληση. Τούτου λεχθέντος συμφωνώ ότι πρέπει να εξεταστούν τα κριτήρια. Όμως θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας. Εντός της Ευρωζώνης θέλω να πω ότι έχουμε σύμφωνο ανάπτυξης και σταθερότητας που όπως ξέρετε είναι πιο βαριά τα, οι κυρώσεις εντός Ευρωζώνης που επιβάλλονται από ό,τι εκτός που μπορούν να επιβληθούν κατόπιν προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. πρέπει να δούμε στην Ευρωζώνη ποιο είναι το κόστος αναμονάδα από τους φορείς ανταγωνιστικότητας, ακόμα και αν δεν υπάρχει πλαίσιο όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αλλά είναι σημαντικό αυτό για την εύρυθμη λειτουργία και ζητούμε αένα διαθωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις. Ακόμα και αν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά διότι είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία ιασδήποτε οικονομία πολλό μάλλον δε τη Ευρωζώνης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Ε, μάλιστα τα είπαμε όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανασυνεδριάζουμε στις 9 το πρωί και έχουμε την Επίτροπο Κρούζ και τον Ζαν claude Juncker που θα μας κυριευτούν. Ευχαριστώ τους διερμηνείς που παρέμειναν. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.